Uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έχω την δυνατότητα να προεδρεύσω στην πιο σημαντική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Εξωτερικών ε, Υποθέσεων αλλά ε, ο Έλμαρ Μπρόκ θα έρθει σε 10 λεφτά και πρότεινα ο κύριος ε, Μπούζεκ να προεδρεύσει που είναι κάποιες μέρες πιο μεγάλο στην ηλικία από μένα αλλά μου είπαν ότι είμαι ο πρεσβύτερος από πλευρά θητείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγαπητέ Τζέρτζι, οπότε σας καλωσορίζω όλους. Είναι μεγάλη χαρά για μένα και επίσης με μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, τον οποίο σας παρακαλώ να χειροκροτήσετε θερμότατα. Είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί εδώ είναι και ο πρέσβης σας και εκτιμούμε πολύ την δουλειά του πρεσβευτή σας και ελπίζω και η, αυτού υψηλότσο βασιλιάς να έρθει ε, κάποια μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, για να μην λοιπόν καθυστερώ ε, θα είμαι για λίγα λεπτά στην υπηρεσία της Επιτροπής και μόλις έρθει ο Έλμαρ Μπρόκ θα εγκαταλείψω τη θέση μου και είναι η τελευταία φορά που θα έχω προεδρεύσει σε αυτή την Επιτροπή. Σας παρακαλώ λοιπόν να λάβετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πέτερινγκ. Ε, κύριε Πρόεδρε Πέτεριν και εγώ θα σας απευθύνω το λόγο σαν Πρόεδρο. Έχουμε 10 ε, λεπτά μέχρι να έρθει ο κύριος Μπροκ και θα έχουμε τελειώσει με τα σημαντικά και τότε θα είμαστε απλώς στις απαντήσεις των ερωτήσεων. Αλλά με τιμάει πάρα πολύ ότι είμαι εδώ σε αυτή την ε, επιτροπή μετά από δύο χρόνια που είχα είχα απευθύνει λίγα λόγια και είχα ακούσει τις σοφές συμβουλές σας και ε, σας βλέπω όλους να δείχνετε νέοι και ωραίοι και ε, βασιζόμαστε στην εμπειρία σας στις σχέσεις μας με την Ευρώπη σχετικά με τις ε, ε, προκλήσεις τις οποίες πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι η βοήθειά σας ε, είναι ανεκτήμητη και θέλω να σας πω ότι από όταν είχα έρθει τελευταία φορά, δηλαδή στα δύο χρόνια που πέρασαν έκτοτε, από πλευράς ε, σχέσεων ε, Ευρώπης και ε, η Ορδανίας πέρασαν μερικά ορόσημα και η Ορδανία επέτυχε πριν από 1,5 χρόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα καθεστώς για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ε, που αντικατοπτρίζει τις εξαιρετικές ε, σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας και μία δέσμευση από την Ιορδανία την οποία εκπροσωπώ εδώ να ακολουθήσει την ε, οδό της ενισχύσεως και συσφίξεως των σχέσεων μεταξύ μας και πριν ε, από μερικές ε, εβδομάδες είχαμε στην Ερυθρά Θάλασσα την συνεδρίαση της κοινή Task Force κάτι που θα θυμούνται για χρόνια οι Ορδανοί διότι αυτή η δύναμη στηρίζει τον βασιλιά όσο ηγείται του προγράμματος ε, εξυγχρονισμού στην Ιορδανία και αποτελεί μία τομή ε, ε, από όλου τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, τα κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις πολιτικές ομάδες, τα κόμματα, την κοινωνία των πολιτών, δημοσιογράφους αφούς δηλαδή ήρθαν ε, εκπρόσωποι όλων των ε, ε, κοινωνικών εταίρων, συναντήθηκαν με τους Ιορδανούς, είχαμε και επιχειρηματίες από την Ευρώπη που συνάντησαν τους απλούς πολίτες της Ιορδανίας και όλα αυτά κατέληξαν εις ένα μεγαλοπρεπές γεύμα που προσέφερε ο βασιλέας, ε, ο βασιλιάς και ε, όχι μόνο συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και της Ιορδανίας αλλά στηρίζει και την πίστη του, της μεγαλειότητος του, αυτού μεγαλειότητος ή στην Ευρώπη ε, σε μια ε, περίοδο μεγάλης αστάθειας και για τους Ιορδανούς ήταν πολύ σημαντικό την ε, αμετάκλητη πορεία προς την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Τώρα ε, εορτάζουμε τη δεκαετία της συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ Ορδανίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τόσα πολλά έχουν συμβεί, τόσες πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί που πραγματικά μιλάμε για ε, μια ιστορία επιτυχιών και είμαστε και δεσμευόμαστε ακόμη περισσότερο ε, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτή τη σχέση. Πρέπει να σας πω ότι με την Ευρώπη δεν είναι απλώς μία φιλία, είναι μία πραγματική ε, ε, εταιρική σχέση μια συνεργασία που δείχνει πως μια χώρα από ένα διαφορετικό μέρος του κόσμου που τους τελευταίους 18-19 μήνες είχαμε πολλές ταραχές μπορεί να εφαρμόσει μια πολιτική και να συσφίξει τις σχέσεις της με την Ευρώπη. Ε, χάρηκα διότι υπεδέχθη την ε, Λέδη Άστον στην Ιορδανία για να ε, επισφραγίσει τη φιλία μεταξύ της Ιορδανίας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρώπη και έχοντας ε, ε, διαπιστώσει ότι υπάρχει μία πολιτική στήριξη αλλά και στήριξη για να αντιμετωπίσουμε τις ε, οικονομικές προκλήσεις και ε, ανάπτυξη διαφόρων προγραμμάτων, προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, εξετάσαμε ε, συνεκτικά όλα τα προγράμματα μεταφορών, παραδείγματος χάρη, που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν την Ιορδανία και να βελτιώσουν και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη χώρα μου και να μας βοηθήσουν να επιλύσουμε και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις τις οποίες ε, ε, ε, συναντούμε και δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει επέμβαση όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την περιοχή και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εταιρική σχέση. Πλέον αυτού θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς τις Βρυξέλλες και αλλού και θέλω να σας πω ότι ε, εκτιμούμε την ε, συνεργασία για την ελεύθερη διακίνηση και ε, τις εμπορικές σχέσεις και δεν θέλω να σας κουράσω με πληροφορίες τις οποίες έχετε ήδη διότι η Επιτροπή σας είναι μία από τις πλέον διακεκριμένες διεθνώς και γι' αυτό θα θεωρήσω ότι δεν μιλώ μόνο σε άτομα που είναι πολύ πιο έξυπνα από μένα αλλά είναι και πολύ καλά πληροφορημένα. Τον Οκτώβριο του 2011 όταν ήμουν στην Ερυθρά Θάλασσα ή στο Οικονομικό Φόρουμ που οργανώνουμε κάθε χρόνο στην Ιορδανία Είδα ότι ε, υπήρχαν ορισμένα γεωστρατηγικά σενάρια για το 2012 και ε, υπήρχε ε, άμεση τηλεοπτική αναμετάδοση και ο κύριος Μούσα ήταν εκεί που είναι τώρα υποψήφιος πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Τόνι Μπλερ και άλλοι πολλοί. Και είπα ότι είναι γελίο οποιοδήποτε από εμά να ε, εκπονεί γεωστρατηγικά σενάρια για το 2012 διότι εδώ όταν συνεδριάσαμε το 2010 κανείς δεν φανταζόταν τι θα συνέβαινε το 2011. Οπότε ε, θα πρέπει ε, να α ό,τι και να προγραμματίσουμε μπορεί να πάει στραβά. Διότι το 2011 ήταν μια πολύ ταραγμένη περίοδος για την Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Η Αραβική Άνοιξη όπως τη χαρακτηρίζεται ε, και εγώ προτιμώ να τη θεωρήσω σαν αραβικό ξύπνημα. Δεν είναι ίσως το πρώτο αραβικό ξύπνημα αλλά είναι το ξύπνημα της πλειοψηφίας των πολιτών πολιτών στην περιοχή του κόσμου όπου βρισκόμαστε διότι ε, ο πληθυσμός είναι πλειοψηφικά κάτω των 30 ετών ήταν λοιπόν το ξύπνημα της ε, νεολαίας ε, που επιζητούσε δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, δυνατότητα να συμμετάσχει στην διαμόρφωση του μέλλοντός τους και τη δυνατότητα να έχουν αυτοδιάθεση και αυτοδιοίκηση και αυτά είναι βασικά δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα και γι' αυτό όλοι αυτοί κινήθηκαν και θέλησαν να εισακουστούν. Οπότε στο τέλος οι ηγέτες στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική ε, και εγώ μιλώ εδώ ειλικρινά και άμεσα οι ηγέτες είχαν μία από τρεις επιλογές η πρώτη επιλογή ε, ήταν ότι γνωρίζοντας ότι αναπόφευτα θα υπήρχαν αλλαγές ε, θα έπρεπε είτε να προσαρμοστούν σιγά σιγά ή στις αλλαγές και θεσμικά και γενικά ή να αντισταθούν στην αλλαγή ε, και να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα που είδαμε στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική ή ε, να υπάρξει ε, ραγδαία αντίδραση και ο, η αυτού μεγαλειώτης ο βασιλέας μας είχε προλάβει αυτές τις εξελίξεις δεν ήταν ευχολόγιο αλλά ε, γεγονός. Μπορώ να συνεχίσω κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τι σας έλεγα Αυτά είναι γεγονότα για τα οποία είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Το γεγονός ότι στην Ιορδανία όπως περιέγραψε η Κάθη Άστον υπήρξε αλλαγή προληπτική χωρίς χαός με μεταρρυθμίσεις πολιτικές τις οποίες προετοιμάζαμε από πολλά χρόνια πολλές φορές όπως είπε ο βασιλιάς κάναμε ένα βήμα μπρο και δύο πίσω υπήρχαν απρόβλεπτα γεγονότα αλλά η δέσμευσή μας ήταν αμετάκλητη και εις ε, την χώρα μας που είναι στην καρδιά της Μέσης Ανατολής το σταυροδρόμι ε, αυτό μεταξύ νέων και παλαιών πολιτισμών ε, σε ένα σημείο που όπου υπήρχαν διάφορες αλλαγές και βεβαίως μία γέφυρα μεταξύ βορρά και ε, νότου. Οπότε οι άνθρωποι λένε γιατί κάνουμε ένα βήμα μπρο και δύο πίσω. Ποια είναι τα γεγονότα πέραν ε, των δυνατοτήτων σας και γιατί ε, η, η περιοχή ε, επεμβαίνει και επιβάλλει το τι πρέπει να γίνει. Ε, είχαμε τρεις πολέμους, οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Είχαμε ε, τον πόλεμο στο Ιράκ, τον πόλεμο στο Λίβανο, τον πόλεμο στη Γάζα. Ε, σκεφτείτε τι πόροι χρειάστηκαν και υπήρχαν αυτά τα γεγονότα τα οποία ήταν εκτός του ελέγχου μας και η διάσταση ε, ε, των σχέσεων ε, Ισραήλ και Παλαιστίνης και οι πολιτικές αλλαγές στις διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων και στην Ιορδανία που είναι εμπλεκόμενο μέρος γιατί και εμείς αντιμετωπίζουμε στην Ιορδανία προκλήσεις οικονομικές, ε, οικονομικές δυσχέρειες και τέλος πρέπει να μην ξεχνάμε ότι εισάγουμε 96% της ενεργείας μας. Μόνο το 2011 χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε ε, δύο δύσκολα γεγονότα. Πρώτον, μία αύξηση κατά 50 δολάρια το βαρέλι ε, ε, μεταξύ το φθινόπωρο του 2010 μέχρι την άνοιξη του 2011 στο πετρέλαιο που επιβάρυνε πάρα πολύ τον προπολογισμό της Ιορδανίας και για τη χώρα μας ήταν ένα βαρύ πλήγμα και το δεύτερο βαρύ πλήγμα ήταν ε, η ε, διακοπή της παροχής αερίου από την Αίγυπτο στην στην Ιορδανία διότι 12 φορές ανατινάχτηκε ο αγωγός και ε, κάθε ημέρα διακομή, διακοπής οδηγούσε ε, σε, σε μια επιπλέον επιβάρυνση για την Ιορδανία που κόστιζε 5 εκατομμύρια δολάρια. Για κάντε τα μαθηματικά και θα δείτε αν τα υπολογίσετε πόσα βγαίνουν. Και σε όλα αυτά έπρεπε να υπάρξει και ένα πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έπρεπε να προωθεί λαμβάνοντα λαμβάνοντας υπόψη όσα συνέβαιναν και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι εξελίξεις στην Ιορδανία ήταν ή επαναστατικές ή εξελικτικές. Είδαμε λοιπόν δύο εξελίξεις επαναστατικές με κάποια βία αλλά χωρίς ανεξέλεγκτες πορείες όπως είδαμε στην Ισία και στην Αίγυπτο και ε, βλέπουμε ότι ε, στην περιοχή υπάρχουν ακόμη γεγονότα εν εξελίξη. Ε, είδαμε τι έγινε στην Λιβύη, τι έγινε στην Ιεμένη, τι γίνεται ακόμη στη Συρία. Οπότε στη χώρα μου η αυτού μεγαλειώτης πιστεύει στην δύναμη και στις δυνατότητες της νεολαίας και αυτό οδήγησε στο ότι η χώρα μας κοίταξε προς τα εμπρός και έδωσε στους νέους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το μέλλον. Τι κάναμε λοιπόν το 2011, κοιτάξαμε την αρχή του αραβικού ξυπνήματος και είπε είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε θετικά τις εξελίξεις αυτές, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ένα βήμα μπρος και πίσω δυστυχώς γιατί σας είπα ότι πολλά από τα γεγονότα είναι πέραν του ελέγχου μας αλλά οι εξελίξεις είναι προφανείς και απτές. Δημιουργήσαμε λοιπόν μία επιτροπή κοινωνικού διαλόγου του 2011 με δύο κεφάλαια. Καταρχήν να υπάρξει ε, εκλογικός νόμος και να υπάρχει ένας νόμος για τα πολιτικά κόμματα. Ο Βασιλιάς δεν είπε ότι αυτά είναι μία διαδικασία η οποία θα είναι ατέρμον. Είπε ότι θέλουμε μία κυβέρνηση η οποία θα εκλέγεται από το Κοινοβούλιο που θα εκπροσωπεί το πλειοψηφικό κόμμα στο Κοινοβούλιο και για να επιτευχθεί αυτό έπρεπε να υπάρχει ένας σωστός εκλογικός νόμος και ένας πολιτικός νόμος που να ρυθμίζει τα θέματα των πολιτικών κομμάτων. Ε, κόμματα τα οποία υπάρχουν εδώ και δεκαετίες και εκτός από ένα-δύο τα οποία είναι οργανωμένα με μια σωστή δομή πολιτική και κοινωνική ε, αλλά είναι προσωποπαγή ή είναι ε, ε, κόμματα τα οποία εμφανίζονται και μετά εξαφανίζονται. Έπρεπε λοιπόν να αλλάξει όλη η φιλοσοφία να μπορέσουμε να έχουμε μία παιδεία για τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά κόμματα αυτά να εκλέγονται στο Κοινοβούλιο διότι πιστεύετε σε αυτά τα οποία εκπροσωπεύουν και η Εθνική Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της εντός των τριών μηνών που είχε θέσει σαν χρονοδιάγραμμα και χωρίς ε, αντιρρήσεις. Δηλαδή είπαμε έπρεπε να αλλάξουμε ορισμένα άρθρα στο Σύνταγμα του 1952 και γι' αυτό σας είπα ότι προπορεύθηκε ο, η αυτού μεγαλειώτης ο βασιλιάς διότι είπε ότι εγώ δεν θα τροποποιήσω μόνο τις 29 τροπολογίες, θα τροποποιήσω ε, όλο το Σύνταγμα και ε, ε, από τις καταργήσεις 42 από τα 120 άρθρα του Συντάγματος καταλήξαμε σε μία πλήρη αναμόρφωση του νέου Συντάγματος που ψηφίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου και που περιλαμβάνει για πρώτη φορά ίσως στην περιοχή μας μία ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα εποπτεύει τις εκλογές είτε είναι δημοτικές είτε είναι κοινοβουλευτικές και όχι μόνο τις εκλογές αλλά θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μόνη της τις εκλογές. Δηλαδή ε, το θέμα αυτό συζητείται τώρα και η Επιτροπή θα μπορεί να επιλέγει την ημερομηνία των εκλογών και θα ε, εμπλέκει και όλους τους ενδιαφερόμενους της χώρας αυτή τη διαδικασία. Ε, γι' αυτό και σας λέω ότι έχουμε μία προοδευτική εξέλιξη στη χώρα μας και υπάρχει πλέον και ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο ρυθμίζει τα θέματα του συντάγματος πέραν ε, του κοινοβουλευτικού μηχανισμού που ήδη προϋπήρχε. Ολοκληρώσαμε, όπως σας είπα, ένα νομοσχέδιο ε, για τον εκλογικό νόμο, για τα πολιτικά κόμματα, ε, για τις δημοτικές εκλογές. Όλα αυτά συζητούνται τώρα στο Κοινοβούλιο, για τα δικαστήρια και ε, εντός των προσεχών ημερών θα υποβληθεί και το νομοσχέδιο για τις εκλογές και η κυβέρνηση θα έχει επιτύχει αυτό το οποίο επιζητούσε και θα μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε ε, ε, ε, έναν απολογισμό και να προχωρήσουμε σε άλλα θέματα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολιτικές εξελίξεις συμβαδίζουν με τις οικονομικές εξελίξεις όπως και πρέπει. Παρόλο που όπως σας είπα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές προκλήσεις έλλειψη ε, της ασφαλείας και της ειρήνης στην περιοχή είναι μια ανησυχία αλλά η Ορδανία είναι ένας ε, ε, πόλος σταθερότητος και με την απαρχή της Αραβικής Άνοιξης, όπου όλοι αποζητούν τη δικαιοσύνη και την ισότητα, μια ζωή μέσα στην αξιοπρέπεια, με ίσες ευκαιρίες, το ζήτημα της Παλαιστίνης παραμένει το βασικό πρόβλημα δεν μπορεί να υπάρξει πλήρη ε, αραβική άνοιξη, ολοκλήρωση τη διαδικασία αυτή, αν δεν υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρί να επιληθεί η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη. Είναι σαφή η θέση μα προ αυτό το θέμα και είναι γνωστή. Πρέπει να υπάρξει λύση των δύο κρατών. Ανεξάρτητο, βιώσιμο κράτο, ε, ολοκληρωμένο κράτο ε, τη Παλαιστίνη. Βάσει των συνοριακών γραμμών του 67. Το Ισραήλ επίση να είναι ένα κράτο το οποίο να ζει σε συνθήκε ειρήνη και τα δύο κράτη αυτά να συμβιώνουν σε ένα περιβάλλον ασφαλέ για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η προσέγγιση μα στο συγκεκριμένο πρόβλημα και εκεί θα θέλαμε να έχουμε μια προσέγγιση χρήσιμη. Γι' αυτό λοιπόν τι τελευταίες 6-7 εβδομάδες στην Ιορδανία φροντίσαμε να έχουμε σχετικέ συζητήσει. Δεν είμαστε απλώ ένας διαμεσολαβητής, δεν είμαστε απλώ ένας παρατηρητής. Έχουμε κι εμείς συμφέροντα που διακυβεύονται στην συγκεκριμένη αυτή ε, περίπτωση. Υπάρχουν ζητήματα που μας απασχόλουν. Η Ιερουσαλήμ, οι πρόσφυγε, τα σύνορα, το νερό, ε, οι μετανάστε είναι ζητήματα που αφορούν άμεσα και τα πέντε την Ιορδανία. Είμαστε κι εμεί ενδιαφερόμενο μέρο στι συζητήσει. Και όταν προσπαθούμε να φέρουμε κοντά του Ισραηλινού και του Παλαιστινίου, όταν έχουμε διερευνητικέ συζητήσει στην Ιορδανία, αυτό συμβαίνει γιατί πραγματικά είμαστε πεπισμένοι ότι την περασμένη, τον περασμένο 1,5 χρόνο με τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, το αδιέξοδο που αντιμετωπίσαμε δεν χρησιμεύσε σε κανέναν. Το αδιέξοδο αυτό μας απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από την εξέβρεση μια κλίσης, που όλοι όμως την αποζητούμε. Πρέπει λοιπόν να πω ότι είχαμε πέντε γύρους διαβρεμητικών συζητήσεων με τους Παλαιστινίου και τους Ισραηλινούς. Ε, οι συζητήσεις αυτές, ε, μπορώ να σας πω ότι είδα εγώ δηλαδή συμμετέχοντα σε συζητήσει αυτέ, ότι ήταν αρκετά εγκάρδιο το κλίμα, με διάθεση να βρεθεί κάποια λύση, έστω και τεχνοκρατικώς, Είναι μεγάλο όμως το χάσμα μετά τα 6-7 χρόνια κατοχής, μάλλον ε, των ε, τελευταίων εχθροπραξιών και τα τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες κατοχής δεν θα είναι εύκολο να βρεθεί η κατάλληλη λύση, αλλά δεν θέλουμε να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις. Πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έρθουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και πάλι, υπήρξε διαφορετική ερμηνεία της δήλωσης ε, του κουαρτέτου στις 23 Σεπτεμβρίου του 2011 όπου καταδικάστηκε με τη δήλωση αυτή όπου υπήρξε μάλλον ε, συγκεκριμένη καταδίκη μέσα από τη δήλωση και όπου υπήρξε και χρονική προθεσμία. Είπε 30 μέρες για προσκευαστικές ομιλίες στο κουαρτέτο, 90 για τους όρους ασφαλείας και άλλες 90 για να υπάρξουν πρόοδο για τα δύο αυτά ζητήματα και μετά 6-7 μήνε μέχρι να ολοκληρωθεί ένα πρώτο πλαίσιο, μια πρώτη συμφωνία πλαίσιο για όλα. Η ερμηνεία των δύο πλευρών είναι διαφορετική για το πού αρχίζουν οι 90 μέρε, πριν ή μετά τι 26 Οκτωβρίου, λόγου χάρη. Εμένα μου δείχνουν τώρα εδώ ότι η προθεσμία αυτή έχει ήδη εκπνεύσει. Δεν έχω άλλο χρόνο μιλίες από ό,τι μου λένε. Αλλά να πω ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι σημαντικό στοιχείο για όλους και θα φέρει ηρεμία και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Είναι παγκόσμιο το ζήτημα και έχει παγκόσμιε διακλαδώσει. Θέλω να μιλήσω και για τη Συρία και μπορώ να σα πω πολύ γρήγορα, συμπερασματικά, ότι ω χώρα που έχει σύνορα με τη Συρία, κοινά σύνορα με τη Συρία, Συρία μα απασχολούν οι δολοφονίε και το αιματοκύλισμα και οι φρικαλαιότητε που λαμβάνουν χώρα και καθημερινά και θα πρέπει από τη διεθνή κοινότητα να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μια πολιτική λύση. Είναι σαφέ αυτό. Δεν θέλουμε να υπάρξει καμία παρεμβολή που θα αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο την όλη περιοχή. Επίση, ίσω να απαντήσω κάτι το οποίο δεν ανέφερα προηγουμένω, ε, απαντώντα σε κάποια τα ερωτήματά σα. Υπάρχει μια ομάδα που ονομάζεται Φίλοι τη Ιορδανία στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ε, ήθελα να υποθέτω ότι ο καθένα εδώ είναι φίλο τη Ιορδανία. Ε, Και Είμαστε περήφανοι που έχουμε τέτοιου φίλου τη Ιορδανία και είμαστε δεσμευμένοι η φιλία μα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη για όλου σα. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σα προσκλήση σήμερα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας και την ενημέρωση που μας δίδετε. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ θετική και οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να γίνουν με διάφορους σκοπούς. Ελπίζω να επιτύχετε εσείς ε, στη δραστηριότητά σας. Αρχίζει η συζήτηση. Ο Μιχαήλ Κάλα πρώτος. Ευχαριστώ πολύ στα αγγλικά. Και πάλι καλωσορίσατε Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Ε, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ και που ακούμε τις καλές ειδήσει που μας φαίνεται για τη χώρα σας. Όλοι ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κυβέρνησή σας στη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Ξεκαθαρίσατε ότι οι μεταρρυθμίσεις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές θα πρέπει να βγαίνουν χέρι-χέρι. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή θα εξελιχθεί ομαλά και στη χώρα σας. Είμαι και βέβαιος ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σε συνεργασία με τη χώρα σας και την κυβέρνησή σας να βοηθήσει και να συνοδεύσει με θετικό τρόπο αυτή τη διαδικασία. Έχω μια ερώτηση που αφορά πολύ περισσότερο, γιατί είστε και μέλος του Αραβικού Συνδέσμου, ε, εσωτερικά, σε ό,τι αφορά τη Λιβική κρίση. Τι είπα Λιβύη, τη Συρία εννοούσα. Λίμπιαν είπε, του λέει η Ρία. Ναι, ναι, όχι, όχι. Ποια Λιβική, όχι, όχι, τη Συριακή. Ναι. Ε, με ερμηνεύει η Ρία Όμεν εδώ, παρακαθήμενη. Ε, η Συρία και η Λιβύη έχουν κάτι Ι και κάτι Ι, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Αραβικό Σύνδεσμο, επανειλημμένα έχει λάβει θέση για ένα θέμα ενός κράτους μέλους του. Δεν το είχαμε δει αυτό στο παρελθόν επί δεκαετίες Πρόσφατα το βλέπουμε και είναι θετικό, αλλά εκπλήσωμε γιατί αν δει κανείς μια χώρα όπως είναι την Ισία σε μια μεταεπαναστατική περίοδο έχει κάνει μεταρρυθμίσεις, έχει εκλογές, κυβέρνηση, ενώ στη Σαουδική Αραβία δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μεταρρυθμιστική χώρα του κάθε άλλο. Και η δική σας ε, κυβέρνηση ε, συνεχίζει ε, ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό της χώρας. Λοιπόν, βλέπετε αυτές τις τρεις χώρες με πολύ διαφορετική εσωτερική κατάσταση είναι ε, στην ίδια πλευρά και πιέζουν το καθεστώς στη Δαμασκό να μην χρησιμοποιεί βία και να αποσυρθεί ουσιαστικά και να ανοίξει το δρόμο για την αλλαγή στη Συρία. Ποια είναι τα κίνητρα. Τόσο διαφορετικές χώρες, αυτές οι τρεις που σας ανέφερα, έχουν την ίδια θέση. Τι τις οδηγεί σε αυτό. Θα μπορούσατε λίγο να μας εξηγήσετε πώς γίνονται οι συζητήσεις στον Αραβικό Σύνδεσμο. Και άλλη σύντομη ερώτηση για τη Συρία. Έχετε προετοιμαστεί να υποδεχτείτε... Συρία δεν είπα τώρα. Πάλι Λιβύη είπα. Όχι, όχι. Συρία. Είστε έτοιμοι να δεχτείτε πρόσφυγες. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες ξέρουμε ότι προετοιμάζεται η Τουρκία από τη δική της ε, παραμεθόρια περιοχή να δεχτεί πρόσφυγες. Εσείς είστε έτοιμοι, έχετε ήδη υποδεχτεί πρόσφυγες από τη Συρία και προβλέπετε, ας πούμε, οι χριστιανικές μειονότητες έρχονται στη χώρα σας ήδη. Γιατί φοβούμαστε, είδαμε τη μοίρα επιφυλάχθηκε στους ε, Ιρακινούς χριστιανούς. Φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και στη Συρία ε, ενώπιση των ταραχών. Κανείς δεν είναι άχρηστος. Ε, εσύ μπορεί να χρησιμεύσεις ως κακό παράδειγμα λόγω του χρόνου αγόρευσης. Λοιπόν, δύο λεπτά για ένα και ενάμιση έχουμε πάρα πολλούς. Ε, κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ που ήρθατε εδώ σήμερα και για τι εξηγήσει σα για τι εσωτερικέ μεταρρυθμίσει. Ελπίζω να πετύχουν, διότι ακούω πολύ θλιβερέ ε, ειδήσει από την ελευθερία στον κόσμο για το 2012 και το ότι αντίκτυπο υπάρχει από την Αραβική Άνοιξη. Η Ορδανία δεν έχει και πολύ καλή θέση ω προ τι ελευθερίε των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λίγο παραπάνω από από το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Ε, αυτό λοιπόν που μας είπατε, η όλη περιγραφή σας, μεταρρυθμίσεις ελπίζω να πετύχουν. Εκτιμούμε βεβαίω το ρόλο που έχετε διαδραματίσει διεθνώ και εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό που είπατε χθε, ότι η Ορδανία θα προσχωρήσει στην Σύμβαση για τα Βιολογικά και Χημικά Όπλα και στο NPT. στη Σύμβαση για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Όμω, ε, προκειμένου να γίνουν όλα αυτά, τι ε, συστάσει θα μπορούσατε να απευθύνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ να μεταχειριστεί την περίπτωση του Ιράν. Επίση, για την περίπτωση τη Συρία. Εκτιμούμε ιδιαίτερω την στήριξη που έχετε προσφέρει στο λαό τη Συρία. Αλλά θα θέλαμε και τι απόψει σα για τον κατακαιρματισμό που επικρατεί στη χώρα αυτή. Η αντιπολίτευση πώ μπορεί να ενισχυθεί, να ξεπεράσει αυτόν τον κατακαιρματισμό που είναι προφανώ ε, εμπόδιο για το μέλλον. Η Ιορδανία θα ήταν πρόθυμη εντός της, ε, του Αραβικού Συνδέσμου να ζητήσει την παραπομπή του Πρόεδρου Ασάντ στο Διεθνές Δικαστήριο και άλλων για την η συμπεριφορά τους και τη βία εκστρατεία τους κατά του λαού της Συρίας. Η κυρία Νέιτς. Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, Υπουργέ, εξ ονόματος ε, της ομάδας των φιλελευθέρων σας καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχασα το πρώτο τμήμα και ζητώ συγγνώμη και ίσως η ερώτησή μου να έχει ήδη απαντηθεί. Και πάλι θα σας ζητήσω συγγνώμη. Έχω τις εξής δύο ερωτήσεις. Ανέκαθεν θαύμαζα τον τρόπο με τον οποίο ε, συμμετείχαν ε, και το ρόλο που έπαιζαν οι βασίλισσες στην Ιορδανία, στην οικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτόματα με φέρνει αυτό στην ερώτηση τι ρόλο διαδραματίζουν οι γυναίκες στην Ιορδανία ε, στις μεταρρυθμίσεις σήμερα και υπάρχουν τίποτα ειδικέ διατάξεις για περισσότερη ισότητα των φίλων στην Ιορδανία. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. ερώτηση δεύτερη έχει σχέση με τη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση ε, Παλαιστίνης-Ισραήλ. Θα ήθελα τις απόψεις σας, ή δυνατόν, για την κατάσταση των πραγμάτων και πώς έχει η συμφιλίωση ή η μη συμφιλίωση μεταξύ της Χαμάς και της Φατάχ. Και αυτό πώς επηρεάζει τις συνευτικές συνομιλίες. Ευχαριστώ δεν Η κυρία Μπρέπολς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα, ε, θα ήθελα και εγώ εξ ονόματος των Πρασίνων και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας να καλωσορίσω τον Υπουργό και να τον ευχαριστήσω για την εκτενέστατη εισαγωγή και παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα του. Μπορείτε σας παρακαλώ να διευκρινίσετε λίγο περισσότερο για μας για το τι σημαίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις για τους Παλαιστινίους που είναι πάνω από 2 εκατομμύρια η ε, Παλαιστίνη από τη Δυτική Όχθη λεγόμενη που ε, σε πολλές ε, δομές σήμερα αποκλείεται η συμμετοχή τους και στις κρατικές υπηρεσίες και αλλού σε αντίθεση με εκείνους που είναι από την Ανατολική Όχθη, Ε, η Ορδανία τη στηρίζουμε και εμείς με 200 εκατομμύρια, αλλά για το 2011 η Σαουδική Αραβία έχει δώσει πάνω από ένα δις εκατομμύριο ευρώ στην Ιορδανία. Αυτή η στήριξη συνδέεται με όρους και προϋποθέσεις, ε, οικονομική βοήθεια που έρχεται από διάφορες πλευρές και στόχος είναι πραγματικά να προωθήσει τη δημοκρατία στην Ιορδανία. Άλλη ερώτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το είπε και η κυρία Νέιτς. Η χώρα σας χαίρει φήμης πολύ καλύτερης ε, από πολλές γειτονικές χώρες σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ε, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα λοιπά. Ε, πρόσφατα προσχωρήσατε σε μια σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστήριων. Αλλά πέρυσι σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου έπεσε από την 120η θέση στην 128η. Ε, πρόσφατα είχαμε τον πρέσβη κύριο Αντάμι του Αραβικού Συνδέσμου στην αντιπροσωπεία για το Μασρέκ και μας είπε ότι γίνονται μεγάλες ε, συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις στον Αραβικό Σύνδεσμο και πώς επηρεάζουν ε, οι μεταρρυθμίσεις της Ιορδανίας τις συζητήσεις που γίνονται ε, στον Αραβικό Σύνδεσμο. Ο Σερ Ρόμπερτ Άτκινς. Υπουργέ, έρχεστε από μια χώρα που είναι πρότυπο υγείας, ευρωστίας και κοινή λογική ε, στο αδιέξοδο που βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Και η αυτού μεγαλειώτη ε, το εκπροσωπεί αυτό και η Υπουργή. Ε, έχω τα εξή ερωτήματα τώρα. εφού η Χαμά έχει εγκαταλείψει τη Δαμασκό και υπάρχει την τρέλα να παραμένει στη Συρία, γιατί η Ουρδανία δεν προσφέρει έδρα στα επιτελεία της Χαμάς. θα ήταν μια απαραίτητη μερίδα ανθρώπων αυτοί με του οποίου θα θέλαμε να συνομιλήσουμε για να επιληθούν τα ζητήματα τη Μέση Ανατολή. Και λαμβάνοντα αφορμή από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, η ε, γύτητα μεταξύ των ε, Χαμά και Φατάχ και όσα δήλωσε ο Υπουργό Υπουργός ε, το κατά πόσον θα εφαρμόζουν τον κανόνα του Διέρνη και Βασίλευε. Αυτά ε, ω σύγκληση θα μπορούσε να εξυπηρετήσουν του σκοπού μα. Και κατά τρίτον, οι σχέσει μεταξύ Ιρδανία και Ισραήλ σε τι φάση βρίσκονται. Υπάρχει μια δεξιά κυβέρνηση, δεξιά ε, παράτα... παράταξη κυβέρνηση στο Ισραήλ. Αυτό κατά πόσον θα μπορούσε να πλήττει τις σχέσεις ε, Ισραήλ και Ιορδανίας κατά πόσο θα μπορούσε να τι υποβαθμίζει. Και τέλο, πιστεύετε, Υπουργέ, ότι το κουαρτέτο είναι ίσω μια υπερβολή, διότι εμεί ε, πληρώνουμε ένα πολύ, καταβάλουμε ένα πολύ σοβαρό κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε αυτό το έργο. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση με το έργο του κουαρτέτου, το οποίο δεν φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω από ένα πρόσχημα για τον κύριο Μπλερ για να προβάλλεται στην, ε, ως ευεργέτης της Μέσης Ανατολής. Εάν δεν αν ισχύει λοιπόν κάτι τέτοιο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να λειτουργήσει το όλο σύστημα. Κύριε Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε, Υπουργέ. Εδώ είμαι. Καλώ ορίσατε, Υπουργέ. Και από την ομάδα μου σα καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα είναι ο κοινό παρονομαστή τη αραβική αφύπνιση, όπω την ονομάσατε, ή τη άνοιξη είναι ότι έφτασαν στην εξουσία Ισλαμικά κόμματα παντού. Στις δικές σας μεταρρυθμίσεις στη χώρα σας προβλέπετε εκλογές και σύντομα. Και από ό,τι φαίνεται και στην Ιορδανία γίνουν εκλογές, μπορεί το Ισλαμικό κόμμα να είναι πρώτο κόμμα. Ισλαμιστικό. Και η Συριακή κρίση που έχει και οικονομικές και στρατηγικές επιπτώσεις. 73.000 ε, πρόσφυγες μπορείτε να δεχτείτε και σας τιμά αυτό. Πιστεύετε ότι αν γίνουν εκλογές μετά τις μεταρρυθμίσεις και στην Ιορδανία μπορεί να βγει πρώτο κόμμα ένα Ισλαμικό κόμμα. Κάτι άλλο τώρα θα ήθελα να ρωτήσω. Ποια είναι η άποψη της κυβέρνησής σας σε σχέση με τις ε, εξαγγελίες που έκανε το κράτος του Ισραήλ για στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν. Θα με ενδιαφέρει η απόψή σας. Και τέλος, το λεγόμενο Εθνικό Ιορδανικό Συμβούλιο ξέρετε ότι έδωσε συνέντευξη τύπου ε, στην Ουάσιγκτον. Είναι μη αναγνωρισμένη αντιπολίτευση και ε, κάνει λόγο για οικονομικές ατασταλίες στη διεθνή οικονομική βοήθεια. Θα θέλετε παρακαλώ να μας το σχολιάσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι einmal. Thank you very much. I mean... Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις και παρεμβάσεις και ουσιαστικά τα ζητήματα θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ καλύτερα. Ε, τα εσωτερικά κίνητρα του Αραβικού Συνδέσμου. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, είναι ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος δίνει το ύφο και προσπαθεί να ε, ρυθμίσει τα των Αράβων εντός του αραβικού οίκου. Εσείς ε, ε στην ερώτησή σας, μια σύγχυση οδηγηθήκατε ε, ανάμεσα στη Λιβύη και τη Συρία, κύριε Γκάλερ, γιατί ε, το 2011 είχε ε, πολύ στεναρή και προχωρημένη θέση ο Αραβικός Σύνδεσμος για τη Λιβύη. Και εκεί βασίστηκε η διεθνής κοινότητα όταν ελήφθη η απόφαση το ψήφισμα 17, 1973 συγγνώμη, και η απαγόρευση υπέρπτυσης. Βοήθησε πολύ λοιπόν ο Αραβικός Σύνδεσμος γιατί έδωσε τον τόνο, το ύφος και τη θέση που χρειάζεται για τη διεθνή κοινότητα και που χρειάστηκε για να προχωρήσει. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη του Αραβικού Συνδέσμου ε, δεν μπορούν να πούν ότι τους επιβλήθη έξωθεν η παρέμβαση και επέμβαση. Ε, στη Συρία η κατάσταση είναι διαφορετική είναι διαφορετική από τη Λιβύη, είναι πιο περίπλοκη. Είχαμε 8-9 συνεδριάσεις στου τελευταιου 6 6-7 μήνε Υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου και περάσαμε ψήφισμα μετά από ψήφισμα. Και μάλιστα ζητήσαμε να πάμε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει το αραβικό σχέδιο για πολιτική λύση στο συριακό πρόβλημα. Και είδαμε το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά θα ε, βάλουμε προσπάθειες ως αραβικό Σύνδεσμος να πάμε στη Γενική Συνέλευση και να πετύχουμε ψήφισμα όπερ και γένετο. Είχαμε και τη ε, συνεδρίαση των φίλων της, ε, της Συρίας στην την Ισία. Είναι μια χώρα που το τελευταίο διάστημα πέρασε τόσες αλλαγές και ήταν και αυτό συμβολικό και σημαντικό. Λοιπόν, ο αραβικό σύνδεσμο μπορεί να έχει διάφορα χαρακτηριστικά στου κόλπου του και οι χώρε. Εγώ δεν είμαι σε θέση τώρα να κρίνω ε, οποιαδήποτε χώρα. Μπορώ να μιλήσω για τη χώρα μου. Ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο κοινό παρονομαστή είναι ότι θέλουμε πολιτική λύση και όχι εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Ούτε διχασμό, ούτε συμβιβασμούς ως προς την εδαφική της ακαιρεότητα. Είναι πολύ περίπλοκη η περίπτωση της Συρίας. Ίσως απαντώ και σε άλλες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Συριακής κοινωνίας ε, και τους πρόσφυγες. Και δημογραφικά ο κοινωνικός ιστός είναι τέτοιος ε, που έχει πάρα πολλές προελεύσεις και διαφορετικές ρίζες. Έχουμε χριστιανούς, ε, ε, Άραβες, Σουνίτες, Κούρδους, ε, Σουνίτες, Αλεβίτες, Σιήτες, Δρούζους κτλ. Πολλές μειονότητες στη Συρία που από κοινού δημιουργούν την πλειοψηφία. Σήμερα οι Αλαουίτες είναι ο πρόεδρος και η οικογένειά του. Και ορισμένοι μπορούν να θεωρούν ότι είναι μια μειονότητα που κυβερνάει την πλειονότητα και πρέπει να διορθωθεί. Στη τελική ανάλυση όμως αυτό που λέμε είναι ότι η αντιπολίτευση δεν ξέρω αν είναι κατακαιρματισμένη όπως ανέφερε κάποιος αξιότιμος βουλευτής. Πάντως ενωμένη δεν είναι. Δεν εμφανίζεται ως συμπαγής ενιαία. Ακόμα και αν διαφορετικές συνιστώσεις ε, έχουν ε, θεμητό ρόλο. Ε, Ελεύθερο Συριακό στρατό, το Εθνικό Συμβούλιο, διάφοροι ανεξάρτητοι μεμονωμένοι πολίτες καθημερινοί που αγωνίζονται και μάχονται για την αξιοπρέπειά τους και τα δικαιώματά τους και τους πατάσουν ε, βία και ομά. Θα έχουμε κύμα χριστιανών, ρωτήσατε, και για αυτούς προετοιμαζόμαστε. Όχι, για όλους προετοιμαζόμαστε. Είμαστε ευλογημένοι. Ε, στην Ιορδανία συμβιούν αιώνε αρμονικά χριστιανοί και μουσουλμάνοι και η χριστιανική κοινότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο στην κοινωνία μας. Δεν ξέρω αν προετοιμαζόμαστε για ένα συγκεκριμένο είδος προσφύγων. Όχι και απαντώ και στι άλλε ερωτήσει για τους πρόσφυγες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ω προ τα νούμερα που ακούμε. Σήμερα έχουν διαβεί τα σύνορα κάποιοι που αυτό αποκαλούνται ε, πρόσφυγες και είναι 4.000. Αλλά εκείνοι που πέρασαν νόμιμα τα σύνορα, γιατί δεν χρειάζεται θεώρηση διαβατηρίων, επισκέπτες, τουρίστες που έρχονται στην Ιορδανία, ε, έρχονται ε, και παραμένουν για πάντα <laughs> είναι 80.000 αλλά δεν αυτό αποκαλούνται πρόσφυγες ούτε τους κατηγοριοποιούμε ούτε τους κατατάσσουμε ούτε η πατιαρμοστία ε, ούτε έρχονται ως πρόσφυγες αλλά τελικά έχουμε 80.000 μη Ιορδανούς που ζουν στην Ιορδανία και χρησιμοποιούν το νερό μας, την ενέργειά μας, τις ιατρικές υπηρεσίες, ε, την παιδεία κτλ. Βεβαίως και τους καλωσορίζουμε και το ίδιο ισχύει και για τους ε, Ιρακινούς. Μοιραζόμαστε το ειστέρημά μας μαζί τους, αλλά πραγματικά είναι πολύ μεγάλο φορτίο τελικά αυτό για την Ιορδανία. Ωραία. Ε, κυρία Γκόμες, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Εγώ δεν προσπαθώ να φανώ σε αμυντική θέση ότι απολογούμε. Να σας πω τα γεγονότα. Εγώ είμαι υπουργό εξωτερικών, γνωρίζω πολύ καλά τη χώρα μου, επίση γνωρίζω τα όσα γράφονται για τη χώρα μου. Και μην ε, επαφίεστε σε μία πηγή. Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί για να περιγράψει ε, την κατάσταση. Είναι αξιοσέβαστη Human Rights Watch και καλή οργάνωση, αλλά είναι μία πλευρά, ε, μία άποψη. Εσείς λέτε ότι η Ορδανία είναι η χώρα που μαζί με άλλες 10 ή 11 της αραβικής αφύπνισης και οι εξελίξεις ήταν απλές ε, γιατί οι αλλαγές έγιναν χωρίς χάος με την ηγεσία του βασιλέως. Ούτε μια σφαίρα δεν ε, πυροβολήθηκε, δεν, ε, δεν έπεσε ούτε μια βιστολιά, ούτε είχαμε ένα τραυματία ούτε νεκρούς. οι αλλαγές λοιπόν μπορεί να γίνουν με οικονομικό, στο οικονομικό πεδίο και οι μεταρρυθμίσεις. έχουμε και διαδηλώσεις που προστατεύονται από την αστυνομία ε, και αν δείτε τις πρόσφατες ε, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και το νέο σύνταγμα, ελπίζω ο πρέσβης μας να σας στείλει αντίτυπα σε όλους, όχι απλώς καταδικάζει τα βασανιστήρια, αλλά και τα στοιχεία που αποσπώνται ε, μετά ε, από βασανιστήρια, τις ομολογίες δηλαδή. Ήμουν και υπουργό ε, ενημέρωσης προηγουμένως πριν γίνω υπουργό εξωτερικών, ήρθε Human Rights Watch και τους είπαμε, ελάτε, μας είπαν θέλουν να δούμε τις φυλακές, να πάτε σε όλες τις φυλακές και να φύγετε και να μην μας πείτε τίποτα. Τέσσερα-πέντε χρόνια πέρασαν και επισκέφθηκαν και τα κέντρα αποκατάστασης και τις φυλακές. Και βρήκαν έναν αστυνομικό που έκανε ε, κατάχρηση εξουσίας γιατί ε, είχε κακοποιήσει, ε, σωματικά είχε προπυλακίσει ένα κρατούμενο, πολύ λάθος και κακό, με μονομένη περίπτωση και απομακρύθηκε. Αλλά δεν υπτίθεται θέμα βασανιστήριο στην Ιορδανία και το γνωρίζει η Human Rights Watch, το παρατηρητήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και κάθε φορά που έρχονται και μας ζητούν πρόσβαση στις φυλακές και οπουδήποτε θέλουν, ε, τους ε, τη ε, παρέχουμε. Δεν λέω ότι είμαστε αλάθητοι. Μπορεί να ξεφύγει κάποιος μια μεμονωμένη συμπεριφορά η οποία απομονώνεται αυτή τη στιγμή διαπιστωθεί. Πραγματικά ταπεινά σας συνιστώ να μην επαφίεστε στα όσα λέει Human Rights Watch. Α, Freedom House, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Εν πάση περιπτώσει, τι λέει μια οργάνωση. Για το Ιράν, ρωτήσατε. Μην νομίζει Human Rights Watch ότι τους ε, στοχοποιώ. Σέβομαι ε, την κάθε οργάνωση, αλλά πραγματικά ας έρθουν να δουν τι κάνουμε στη χώρα και τι λέει το νέο σύνταγμα. Για το Ιράν. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε χώρα έχει δικαίωμα να έχει ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Βεβαίως υπάρχει ένταση και πίεση σε ό,τι αφορά το ιρανικό ζήτημα, την ασφάλεια των κρατών του Περσικού κόλπου και ε, την ανάμειξη στα εσωτερικά μιας χώρας. Θα πρέπει να το δούμε αυτό μέσω διαλόγου, ε, άπαξ διαπαντός και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Εμείς ανησυχούμε ότι αν το Ιράν θελήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή, αλλά θα οδηγήσει και σε κούρσα εξοπλισμού ε, πυρηνικών ε, στην περιοχή και τελικά ε, δεν θα έχουμε τη Μέση Ανατολή που εμείς επιθυμούμε που είναι χωρίς πυρηνικά όπλα. Για την αντιπολίτευση στη Συρία απάντησα. Οι γυναίκες στην Ορδανία διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία το παράδειγμα το απόλυτο και τέλειο είναι η Βασίλισσα, αλλά αν δείτε τις γυναικές οργανώσεις, τις ε, γυναίκες βουλευτές ε, σε υπουργικές θέσεις και κυρίως στην κοινωνία των πολιτών θα διαπιστώσετε ότι ε, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε και μια Εθνική Επιτροπή πλέον για τα γυναικεία δικαιώματα και βεβαίως στην κοινωνία των πολιτών η συμμετοχή των γυναικών είναι ε, πραγματικά σημείο αναφορά για τις εκλογές, για την κυβέρνηση, για τη συμμετοχή. Συμμετέχουν πάρα πολλοί οι γυναίκες και στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ισότητα των φίλων, όσο μπορούμε το προωθούμε σε ό,τι αφορά τη συμφιλίωση μεταξύ Χαμάς και Φατάχ. Είδα στις 23 του μηνός ε, τον πρόεδρο Αμπάς όταν επέστρεψε από το Κάιρο το ρώτησα τι έγινε μου είπε στη δεύτερη συνεδρίαση είχαν κάποιες διαφορές στην πρώτη συνάντηση είχε επικρατήσει μεγάλη εφορία στη δεύτερη συνάντηση άρχισαν να αναδύονται δυσκολίες και κάποιες ε, προκλήσεις ε, για τις εκλογές, για τη συμμετοχή στην κυβέρνηση ο πρόεδρος Αμπάς λέγει ότι η κυβέρνηση του, τώρα που δέχονται να είναι ε, πρωθυπουργός, ε, θα είναι μη κομματικοί, τεχνοκράτες, ανεξάρτητοι, υπερκομματικοί και θα εφαρμόζουν τη δική του πολιτική. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν το Ισραήλ, να δεχτούν ε, τις αρχές της τετραμερούς του κουαρτέτου. Από ό,τι φαίνεται είναι σε ήρεμα νερά αυτή η υπόθεση, αλλά ο πρόεδρος Αμπάς είπε ότι η συμφιλίωση δεν ε, αντιτίθεται στη συνέχιση των ηρευτικών συνομιλιών. Θέλει ο Παλαιστινιακός οίκος να είναι ενωμένο, να είναι ενιαίος για να μπορεί να ε, προχωρήσει και στις υπόλοιπε ενέργειες στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Οι μεταρρυθμίσεις τώρα. Και είπατε ότι οι Παλαιστίνοι στην Ιορδανία εφίστανται διακρίσεις. Δεν θα συμφωνούσα οι Ορδανοί Παλαιστινιακής καταγωγής είναι βασικό στοιχείο της κοινωνίας μας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τους περιγράφουμε ως δεχόμενους διακρίσεις, έτσι με ένα γενικό αφορισμό. Σημειώνω την ανησυχία σας. Σε τελική ανάλυση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το εξής βασικό. Η Ορδανία είναι ένα χωνευτήρι Έχουμε ε, από την Ανατολική Όχθη του ε, Ιορδάνη, Ιορδανούς και Παλαιστινίους από τη Διοικητική Όχθη που είναι και πρόσφυγες και μη πρόσφυγες. 1,9 εκατομμύρια είναι οι μη εγγεγραμμένοι ε, Παλαιστίνοι πρόσφυγες που έχουν ιορδανικό διαβατήριο και υπηκότητα. Αυτό δεν τους αποκλεί όμως από τη δυνατότητα να επιλέξουν όταν έρθει η ώρα το κράτος τους και να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Και αυτό είναι ένα θέμα του τελικού καθεστώτος διαπραγμάτευσης Παλαιστινίων-Ισραηλινών. Αλλά μέχρι τότε είναι, οι Ορδανοί πολίτες συγγνώμη, που συμμετέχουν στην κοινωνία, στις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρηματίες, ε, άνδρες και γυναίκες. Και είναι πάρα πολύ λάθος, αν μου επιτρέπετε, να ακούγεται ότι υφίστανται διακρίσεις μπορεί η εκπροσώπησή του στο κοινοβούλιο να έχει κάποια ερωτηματικά. Και αυτού με Γαλλιώτης ο Βασιλέας επίσημα δήλωσε ότι ε, στις νέες εκλογές η Βουλή θα αντανακλά ε, τη δημογραφική πραγματικότητα ίσως με τρόπο πιο ακριβή. Αυτά θα πρέπει να γίνουν ε, όντως. Σε ό,τι αφορά την οικονομική βοήθεια προς την Ιορδανία αν ε, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις ανάλογα με την πηγή ε, Σαουδική Αραβία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, καμία προϋπόθεση, ούτε θετική ούτε αρνητική. Κανείς δεν βάζει όρους. Ε, υπάρχει υπεποίθηση ότι η Ορδανία κάνει το σωστό και όπως σας είπα, πέρυσι λάβαμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια από τη Σαουδική Αραβία και κάθε μέρα μας ρωτάνε τι γίνεται με το 1,4 Μα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Σας είπα τι έγινε με το φυσικό αέριο. Να που πήγαν τα λεφτά. Το βασικό πρόβλημα είναι ε, το κόστος της ενέργειας και η ανεργία βεβαίως. Αλλά όταν έχουμε και δύο δισεκατομμύρια ε, δολάρια επιπλέον ακριβώς λόγω της διακοπής παροχής φυσικού αερίου από την Αίγυπτο. Ε, η βοήθεια από τη Σαουδική Αραβία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύτιμη και έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. με μεγάλο θαυμασμό μας αντιμετωπίζουν. Είμαστε η αιχμή του δόρατος των μεταρρυθμίσεων και δεν αντιδρούμε σε κάποιες μεταρρυθμίσεις ή όρους που μας επιβάλλονται. Εδώ έχετε ένα πρόβλημα ε, που ονομάζεται more for more, περισσότερα με αντάλλαγμα περισσότερα. Οι χώρες ε, καταβάλουν προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις ε, ειρηνικές χωρίς να καταφεύγουν στη βία ή σε μη συμβατικές μεθόδους καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης. Κάποιος ρώτησε άλλωστε για την ελευθεροτυπία, εσείς νομίζω. Ελπίζω πραγματικά να βρείτε το χρόνο, μισή ώρα χρειάζεται κάποια στιγμή, τις επόμενες ημέρες, και να μπείτε σε κάποιες από τις ιστοσελίδες μας. Πραγματικά σας καλώ να το κάνετε. Μας επιτίθενται, ε, μας... Ε, στριμώχνουν πολλές φορές. Μας εκθέτουν, ε, αλλά πραγματικά θα πρέπει να βασιζόμαστε σε αξιόπιστα στοιχεία ειλικρινή που να επιζητούν ε, την αλήθεια πραγματικά. Αν δείτε πόση ελευθερία ε, έχουμε στην Ιορδανία, ε, ιστοσελίδες, εφημερίδες, ε, μου λέτε τίποτα για το χρόνο πάλι, λοιπόν. Τι έλεγα. Ε, είναι μεγάλη ελευθερία και περισσότερο πολλές φορές από όσοι υπάρχει στην Ευρώπη. Βεβαίως θα πρέπει όλα αυτά να ρυθμίζονται. τώρα, γιατί Χαμάσα θα τη δεχθούμε. Γιατί τα γραφεία ο Χάρετ Μάσερ ε, έχει κάνει επίση επίσκεψη, υπάρχουν ορισμένα στελέχη της Χαμάς που είναι Ορδανοί πολίτες. Γιατί να αρχίσουν να ανοίξουν καινούργια γραφεία, είχαν πριν από το 1999, αλλά τώρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Για τη συμφιλίωση σας μίλησα. Το θέμα δεν είναι εύκολο, αλλά τελικά ο πρόεδρος Αμπάς ε, ε, το προωθεί και το συνεχίζει. Ποιες είναι οι σχέσεις μας με το Ισραήλ. Έχουμε σχέσεις με το Ισραήλ. Ε, στρατηγικά είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ειρήνη με το Ισραήλ. Το 1994 ε, την υπογράψαμε. Ε, θα πρέπει να ωφελήσει και τις δύο πλευρές. Η ιδέα ήταν να έχουμε συνολική ειρήνη. Ακόμα αποσκοπούμε σε αυτό για να έχουμε περιφερειακή συνεργασία και αλληλεγγύη και ευημερία ε, για τους Ισλαμιστές στην κυβέρνηση. Um, Ευχαριστώ. Είπατε αν έχουμε Ισλαμική κυβέρνηση. Δεν ξέρω, θα υπάρξει ένας εκλογικός νόμος, θα υπάρξουν εκλογές και οι εκλογές θα καθορίσουν ποιος πρόκειται να ε, ε, ε, κυβερνήσει σαν κυβέρνηση στην Ιορδανία Ορδανία. Έχουμε μοναρχία αλλά και κοινοβουλευτική και κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε οικοδομήσει και καταργήσει πολλά στο παρελθόν στην Ιορδανία. Ε, έχουμε κόμματα που υφίστανται από 60 έτη ή ορισμένα από τη δεκαετία του 80 και ε, έχουμε και ισλαμιστικό μέτωπο το οποίο ε, αριθμεί 22 από τους 80 ε, βουλευτές του Κοινοβουλίου ε, και η μουσουλμανική αδελφό συνεργάζεται με το σύστημα, είναι μέλος του πολιτικού συστήματος, έχουν κερδίσει εκλογές, έχουν παραμείνει στο Κοινοβούλιο και βλέπετε ότι εμείς δεν έχουμε τις ανατροπές που είδαμε αλλού. Ευχαριστώ κύριος Μπουσουτήλ. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής αλλά είμαι μέλος της ομάδος των φίλων της Ιορδανίας όπως πολλοί συνάδελφοι. Ε, και ε, χωρίς να έχω την άδεια του κυρίου του Σερ Ρόμπερ Άτκινς πρέπει να σας πω ότι ε, θεωρώ ότι η χώρα σας είναι ένας φάρος μέσα σε μια σκοτεινή περιοχή και πολύ μου άρεσε αυτό που είπατε αλλαγή χωρίς χάος και ακριβώς περιγράφει τη διαδικασία την οποία η χώρα σας προωθεί ε, και για να επικροτήσω αυτό που είπατε θα πω αλλαγή χωρίς αιματοχυσία που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στις γειτονικές ε, χώρες και ιδίως στη Συρία και θέλω να τονίσω το θέμα αυτό γιατί η Συρία μας ανησυχεί πάρα πολύ όλους και ναι μεν χαιρετίζουμε την ε, θετική στάση της Αραβικής Λίγκα σας θα ήθελα να ξέρω πώς, του Αραβικού Συνδέσμου θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορεί να σταματήσει άμεσα η αιματοχυσία διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η αιματοχυσία στη Συρία. Επίσης κύριε Υπουργέ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εσείς ε, διαβλέπετε ότι τα θεσμικά όργανα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουν να στηρίξουν τη δημοκρατική εξέλιξη στην χώρα σας και πώς θα οικοδομήσετε αυτά τα οποία ε, ε, προηγουμένως ε, περιγράψατε πώς μπορούμε να σας στηρίξουμε ο, ο κύριος Κράισελ Ντόρφελ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε χαίρομαι που παρουσιάσατε την κατάσταση τώρα στην Συρία υπάρχει μία αντιπαράθεση και θα δούμε ποιος θα είναι τελικά ο συνομιλητής. Εσείς ε, στηρίζετε περισσότερο τον οπλισμένο αγώνα. Ε, πώς τοποθετήστε. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι ότι ε, εμείς είμαστε για την Παλαιστίνη υπέρ της λύσεως δύο κρατών. Αλλά τι θα γίνει με το Ισραήλ, διότι στο τέλος δεν θα μείνει ε, τίποτα από την Παλαιστίνη θα είναι απλούστατα περιφέρειες ε, του Ισραήλ και θα μοιάζει με ένα ε, τυρί ελβετικό με ένα σωρό τρύπες. Ευχαριστώ. Κύριο Κασίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η διαδικασία μεταρρύθμισης του συνταγματό σα ε, και αναβάθμισής του είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για σας, αλλά γιατί και σε άλλες χώρες θα μπορούσε να δοθεί ένα παράδειγμα. Χώρες όπου ε, έχει ολοκληρωθεί ε, αλλά με δύσκολο τρόπο η διαδικασία τη Αραβική Άνοιξη. Επιστρέψαμε από τη Λιβύη από επίσκεψη με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και είδαμε πόσο δύσκολο είναι να εγκαθιδρυθεί και ένα δημοκρατικό καθεστώ. Οι νέοι που συμμετείχαν σε οποιοδήποτε είδο εκλογέ ε, στη Λιβύη είναι τώρα 70 ετών. Δεν υπήρξαν εκλογέ για 42 χρόνια εμπειρία σα, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πολύτιμη σε περιπτώσεις όπως τη Λιβύης. Υπάρχει λοιπόν ε, καμία πρόθεση να τους βοηθήσετε στην όλη διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας και στο πώς να διεξάγουν εκλογές στο μέλλον. Και έπειτα, σε σχέση με τη συνεισφορά σας ε, στην ε, Λιβύη και την επανάσταση εκεί, καθώς και από την εκπαίδευση κάποιων χιλιάδων ε, αστυνομικών. Ε, η ουσία είναι ότι κάποιοι από τους μάχημους αυτούς εκπαιδευόμενους θα επιστρέψουν στις αστυνομικές δυνάμεις της, του κράτους. Όμως το κράτος αυτό ακόμη δεν έχει οργανωθεί. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για, βασική, για το βασικό σκελετό της αστυνομικής δύναμης ε, της χώρας εφόσον τους εκπαιδεύεται ούτως ή άλλως και η υποδομή αυτή λείπει. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ ε, ε, για αυτή την, ε, την ομιλία σας που τόνισε τη συνεργασία, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και είμαι πολύ ευτυχής διότι μας μιλήσατε για τις θετικές εξελίξεις στην χώρα σας. Πώς αξιολογείτε τις μέχρι του προσπάθειες για διαπολιτιστικό διάλογο. Τι μπορούμε να προσφέρουμε επιπλέον στον τομέα αυτό κατά τρόπον ώστε να λάβουμε υπόψη περισσότερο την ποικιλομορφία ε, και ε, τη συλλογική ταυτότητα των αραβικών λαών. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω για την έντιμη αυτή και ειλικρινή παρουσίασή σας ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Όταν οι φίλοι της Ιορδανίας, και έχετε πολλούς φίλους, όπως είπε και ο συνάδελφος Σάιμον, και είχαμε μια ιδιωτική συνομιλία με την αυτομεγαλειότητα των βασιλιά μετά από πρόσκληση στη χώρα σας, η βασική μερίμνα που εκφράσαμε ήταν οι εξελίξει στο Ιράν. Αυτή ήταν η πρώτη μα ανησυχία. Τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ε, αυτό μεγαλειώτη ήταν ε, πολύ ειλικρινή, δεν θα πω τώρα Ποιε ήταν οι λεπτομέρειε του διαλόγου μα, όμω και εκείνο φάνηκε να ανησυχεί ιδιαίτερος. Κατά την άποψή μου, και θα ήθελα να ξέρω αν και εσεί συμμερίζεστε την άποψη αυτή, κατά την άποψή μου, σε αυτή τη χρονική φάση τα πράγματα ουδέποτε υπήρξαν τόσο επικίνδυνα τα τελευταία 50 χρόνια. Αναφερθήκατε, και με αυτό θέλω να κλείσω, στη σημασία και την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην επίλυση του ιστορικού πια προβλήματος μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Νομίζω όμως ότι όλο αυτό θα φανεί πολύ πιο, πολύ λιγότερο σημαντικό σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί στην ευρύτερη γεωγραφική αυτή περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Είμαστε, πιστεύω, στα πρόθυρα εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων και πραγματικά στο κατόφλι στο κατόφλι όχι απλώς ενός ε, τοπικού πολέμου, αλλά μιας ευρύτερης ε, σύγκρουσης σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μία τελευταία ερώτηση. Ε, μήπως μπορείτε να μας ε, συμβουλεύσετε πώς ε, θα μπορέσει να γίνει πιο λειτουργική η σχέση μεταξύ του Αραβικού Συνδέσμου και του Κουαρτέτου ε, των τεσσάρων δυνάμεων διότι θα πρέπει να βρεθεί η σωστή φόρμουλα για να υπάρξει επιτυχία. Μήπως μπορείτε να σχολιάσετε το θέμα αυτό, δηλαδή τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η ευρωπαϊκή πλευρά σαν συμμετέχοντας σε, αυτό το, σε αυτήν την τετραμερή επιτροπή το κουαρτέτο για να μπορέσει να προχωρήσει καλύτερα τα ε, διάφορα θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα πραγματικά ουσιώδη ερωτήματα. Θα ξεκινήσω από εκεί που λογικά τελειώνουν οι σημειώσει μου. Ευχαριστώ για την ερμηνεία αυτή που κάνατε στην αλλαγή χωρί χάο. Αυτή είναι η Ορδανία και αυτή τη δέσμευση έχουμε αναλάβει. Αυτό θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε. Πολλοί είναι εκείνοι που σχολίασαν στι απαρχέ τη Αραβική Άνοιξη ότι εμεί τη διαχείριση του προβλήματο την είχαμε σχεδιάσει πολύ πριν την έναρξη τη Αραβική Άνοιξη. και αυτό φάνηκε με το λαό τη Ορδανία να διαδηλώνει για το ένα το άλλο θέμα αλλά ήδη ξεκίνησαν κάποιε κίνησει στην Ιορδανία πριν την πραγματική αρχή τη Αραβική Άνοιξη. Και μάλιστα οι αστυνομικέ μα δυνάμει προστάτευαν του διαδηλωτέ. Αυτό κάνει τη διαφορά στην Ορδανία. Σα ευχαριστώ για την αναφορά. Λοιπόν, για τη Συρία. Πώ να σταματήσουμε την αιματοχυσία εκεί. Ξέρετε ότι παρακολουθούμε όλοι με φρίκι το τι συμβαίνει καθημερινά. Όχι μόνο εμείς εκείνη την περιοχή, αλλά και στην Ευρώπη και παντού. Καθημερινά. Τα δάκρυα των γυναικών, των παιδιών. Θε... Ε, ήταν ωραία να υπήρχε μια μαγική λύση για να σταματήσει αυτό το δράμα αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια συνολική δέσμευση σε, κάποια περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, μια συνολική δέσμευση όλων μα να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταματήσουν όλα αυτά. Αυτό κάνει και ο αραβικό σύνδεσμο το σχέδιο που είχε παρουσιάσει πριν από λίγου μήνε για να ξεφύγει από αυτό το διέξοδο η Συρία ήταν ένα πολύ καλό σχέδιο. Εμεί προσυπογράψαμε και προσπαθούμε στα πλαίσια του Αραβικού Συνδέσμου να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην υπάρξει εξωτερική στρατιωτική παρέμβαση που θα αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή. Είναι πολύ λεπτομέρειε το πλάνο, το σχέδιο αυτό. Άμεση διακοπή της βίας. Πάυση των δολοφονιών, απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων από τις πόλεις, αστικά κέντρα και να πάνε πίσω στα στρατόπεδά τους, να μπορέσουν αμέσως διεθνείς δυνάμεις, διεθνείς οργανώσεις να έρθουν και να παρακολουθήσουν την κατάσταση, να διευκολύνουν, να ανακουφίσουν ανθρωπιστικά τη χώρα. Διάλογος επίσης με την αντιπολίτευση. Εάν θυμάστε ένα από τα προηγούμενα ψηφίσματα του Αραβικού Συνδέσμου, ήταν από το Κάιρο και τα επιτελεία, τα γενικά επιτελεία του Αραβικού Συνδέσμου να ξεκινήσουν παρατηρητέ προ τη Συρία, αλλά αυτό το αρνήθηκαν οι Σύριοι. Και ε, το τελευταίο σχέδιο του Αραβικού Συνδέσμου που πήγε και στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ και υπήρξε στήριξη ήταν ένα σχέδιο που έλεγε ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια εθνική κυβέρνηση εσωτερική άμεσα Νομίζω αυτή είναι για την ώρα η καλύτερη μας επιλογή. Να συνεχίσουμε να σφυροκοπούμε τα αυτιά των Σύριων με τέτοιες προτάσεις και να καταβάλουμε καθημερινές προσπάθειες. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική λύση εάν δεν προσπαθούμε να αποφύγουμε συνεχώς κάθε δυνατή καινούργια καταστροφή. Ένας από τους συναδέλφους μου πρώην Υπουργό Αραβική χώρα έλεγε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ε, κάνουμε δηλώσει και η αιματοχυσία να συνεχίζεται καθημερινά. Κάποιοι υπουργοί εξωτερικών των αραβικών χωρών του Αραβικού Συνδέσμου δηλαδή πρότειναν μέχρι και το να εξοπλίσουμε του επαναστάτε. Αλλά αυτό δεν είναι μια πολιτική λύση που θα πάψει την αιματοχυσία. Ελπίζουμε ότι οι Συριακέ Αρχέ έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι θαύλο κύκλο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστούν οι δολοφονίε ε, καθημερινά. Κάποια μέρα θα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κατά μέτωπο. Θα πρέπει να συμφιλειωθεί με το λαό. Για την αντιπολίτευση της Συρίας ως ε, συνομιλητή. Αν δείτε τη δήλωση των φίλων της Συρίας και των, του λαού της Συρίας που συναντήθηκαν στην την Ισία. Ακόμη δεν ξέρουμε από ποια αιγίδα να καλύψουμε όλη την αντιπολίτευση της Συρίας. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε διχασμό μεταξύ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης στην ίδια τη χώρα. Πρέπει μεταξύ τους να διοργανωθούν πρώτα. Να υπάρξει μια ενότητα και μετά να αναγνωρίσουμε το Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας ως επίσημο εκπρόσωπο των Συρίων που επιζητούν ειρηνική λύση. Σε ένα πλαίσιο ειρηνικό. Για την πολιτική επικισμού των Ισραηλινών. Συμφωνώ μαζί σας, υπάρχει ε, παντού συνένεση στον κόσμο ότι είναι παράνομη αυτή η τακτική. Οι αλλαγές που συντελούνται είναι καθημερινές. και τα πράγματα φαίνονται να χειροτερεύουν. Διότι όταν συζητά κανεί τι γραμμές του Παλαιστινιακού κράτου, φτάνει πια στα όρια. Αλλά τα πράγματα διαφέρουν από την σκοπιά τη Ιορτανία. Επειδή ακριβώ η πραγματικότητα αυτή είναι καθημερινή, επειδή υπάρχουν παράνομοι επικισμοί και καταβλισμοί στην πράξη, ο μόνο τρόπο να πάυσουν αυτά είναι αν υπάρξει συμφωνία αμέσω για τα σύνορα και την ασφάλεια. Αυτό το λέμε εδώ και ένα-δύο χρόνια. Αν θυμάστε, από το 2009 όταν είχαν έρθει στην ε, αξιότιμη επιτροπή σας. Είχαμε ζητήσει επιτάχυνση της διαδικασίας ε, των συνόρων, αλλά ξεχωριστή αντιμετώπιση τους, να μην τα συνδυάσουμε με όλα τα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Σύντομη, άμεση συμφωνία για τα σύνορα, με ένα περιθώριο τριών ω έξι μηνών. Τότε λέγαμε τρει με έξι μήνε, τώρα λέμε κάτι ανάλογο. Αν κανεί ξέρει τουλάχιστον που βρίσκονται οι συνοριακέ γραμμέ, οποιοδήποτε περνάει και προσπαθεί να χτίσει καταβλισμό από την άλλη μεριά, παραβιάζει τη συμφωνία. Δεν είναι απλώ ότι παραβιάζει μια υποθετική συμφωνία. Πρέπει αυτό να είναι σαφέ, διότι συνεχώ θα ανακοινώνεται η οικοδόμηση καταβλισμών. Ε, και βεβαίω οι διπλωματεύσει δεν θα δίνουν καρπού για τη Λιβύη. Επισκεφτήκαμε και εμεί τη Λιβύη. Και βεβαίω εκτιμούν ιδιαίτερα στο ρόλο που διαδραματίσαμε κατά τη διάρκεια των δύσκολων στιγμών που πέρασαν πέρσι. Μια μεγάλη αντιπροσωπεία τον Οκτώβριο πήγε εκεί και πριν από 15 μέρες το ίδιο με έναν από τους υπουργού μας. Η Λιβύη και η Ιορδανία έχουν πολλά κοινά. Τουλάχιστον στη δική μας τη γεωγραφική ζώνη. Υπάρχουν πολλές πολιτιστικέ ε, ομοιότητες οι Άραβες τον 13ο-14ο αιώνα όταν άρχισαν να μετακινούνται προς τις μας περνώντας από την Βόρεια Αφρική πέρασαν από την Αίγυπτο αλλά μετακινούμενοι με καμήλες χρειάζονταν και γνώσεις τοπογραφίας για να προχωρήσουν. Αγοράζοντας λοιπόν τις καμήλες έφτασαν στη Λιβύη. Αν Δείτε λοιπόν ε, ποιοι κατοικούν στις πόλεις ε, της ε, Λιβύης και σε χωριά της Λιβύης. Είναι πολλοί Βεδουίνοι της Λιβύης που έχουν παρόμοια προφορά με ανθρώπους από το βόρειο τμήμα της Αραβικής Χερσονήσου. Υπάρχουν ομοιότητες λοιπόν στη διαφορά πολιτιστικές, νοοτροπίας μεταξύ Λιβύης και Ιορδανίας. Θέλουμε να του βοηθήσουμε, θέλουμε να του συνδράμουμε και πολλοί κάνουν το λάθο να λένε τη διαδικασία επανοικοδόμηση στη Λιβύη θα πρέπει να γίνει. Μερικέ φορέ δεν μιλάμε καν για επανοικοδόμηση, μιλάμε για οικοδόμηση. Ξεκινούμε από το μηδέν. Δεν είχαν υπουργεία, δεν είχαν σύνταγμα, δεν είχαν διοίκηση, και υπηρεσίε. Πρέπει να του βοηθήσουμε στα πάντα. Βεβαίω, έχουν επιτελέσει σημαντικά επιτεύγματα στην ιατρική λόγω χάρη. Έχουμε ήδη στη Βεγγάζη ένα πειραματικό νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται σε κτίριο ε, ξεχωριστό και εξυπηρετεί ε, χιλιάδες επί χιλιάδων Λίβιους που χρειάζονται αποκατάσταση, θεραπεία αποκατάστασης διότι έπεσαν θύματα ακροτηριασμού. Ναι λοιπόν, στην ανοικοδόμηση, στην ε, υγεία, στην εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων που δεχτήκαμε από στη Συρία λόγω χάρη μπορούμε να διευκολύνουμε τους Λίβιους ε, και με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων τους και με το νομικό τους σύστημα. Χρειάζεται μια προσπάθεια να εξυγχρονιστεί ακόμη και ο τρόπος που προσεγγίζουν τα πράγματα. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα την ερώτησή σας ως προς την πολυμορφία <clears throat> εκτός μικροφώνου ομιλητής στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των χωρών της Αραβικής Άνοιξης, στην Αίγυπτο και το καθεξής. Συμφωνώ. Νομίζω ότι η πολυμορφία είναι αυτό που έχει κάνει τόσο πολύμορφο τον αραβικό κόσμο, αν μπορώ να το πω έτσι. Στην Ιορδανία μιλάμε για ένα χωνευτήρι, όπως το ονομάζω. Έχουμε Αρμένιους, Χριστιανούς, ε, Μουσουλμάνους. Αυτό ισχύει για τη Συρία, το Λίβανο, την Αίγυπτο. Αν και η χώρα είναι πιο ομοιόμορφη, αλλά υπάρχουν και μουσουλμάνοι και χριστιανοί. Η πολιτιστική πολυμορφία θα πρέπει να φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους, όχι να τους ε, χωρίζει. Αυτό είναι η δική μας αντίληψη. Φανταστείτε ότι, ότι ο, κόσμος, ο βασιλιάς μας είναι ο πρωταθλητής αυτό το ζήτημα, διότι κατάφερε στα πλαίσια της κοινοπολιτείας να υπάρξει κοινή μεταχείριση μουσουλμάνων και χριστιανών ε, λόγου χάρη. Θα μπορούσε κανεί λοιπόν να θυμηθεί και το μήνυμα που είχε χρησιμοποιηθεί τότε. Νομίζω ήταν ο πλούτο στην πολυμορφία. Κάτι τέτοιο είχαμε πει τότε. Νομίζω σύντομα θα πρέπει να σιωπήσω, αλλά δηλαδή να ολοκληρώσω. Αλλά όποιο είπε ότι οι εξελίξεις στο Ιράν είναι επικινδυνότερε από ποτέ, νομίζω έχει δίκιο. Εσείς είστε, ναι. Νομίζω οι εντάσεις στον Περσικό κόλπο και οι κόκκινες γραμμές των διαφορών χωρών, είτε από την πλευρά των χωρών τη Δύση ή του Ισραήλ, σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα την ε, παρέμβαση ε, την κατάσταση ασφάλειας του κόλπου είναι πραγματικά ανησυχητικά. Είναι μεγάλη η ένταση και εδώ μπορούμε να δούμε το πλαίσιο σε ένα γενικότερο σκηνικό. Και πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Το κουαρτέτο και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, κύριε Πρόεδρε, ώστε να υπάρχει σκέλος του Αραβικού Συνδέσμου, σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκέλος του Κουαρτέτου, τα οποία να συνεργάζονται. Εσείς ονομάζατε, ε, κύριε στο Κουαρτέτο ένα πρόσχημα για να κάνει ο κύριος Μπλερ τη ζωή του πιο άνετη. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία, όλος ο κόσμος μπορούν μέσω του κουαρτέτου να επιβάλλουν μία λύση σε κάποιου λαού εφόσον δεν το καταφέρνουν μόνοι τους. Αλλά όταν μιλάω για επιβολή λύση, το εννοώ θετικά, όχι κάτι που δεν το επιθυμούν. Ξέρουμε ότι οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλοί επιθυμούν την ειρήνη. Του έχουμε δει να φτάνουν τόσο κοντά στη γραμμή τερματισμού και να μην καταφέρουν να την περάσουν. Θα πρέπει λοιπόν λιγάκι να του καθοδηγήσουμε να τους πούμε ότι και εμείς οι υπόλοιποι στον κόσμο, ως ενδιαφερόμενα μέρη, περιμένουμε επιτέλου την ειρήνη που τόσο έχει λείψει από, τον... από την περιοχή. Εάν δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, να τους βοηθήσουμε. Αυτό θέλουμε και πρέπει νομίζω να τους βοηθήσουμε. Ο κόσμος μας θα ήταν πολύ ασφαλέστερος εάν υπήρχε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, ελπίζω να μην ξεπέρασα πολύ τα όρια του προγράμματος. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ ε, για τα σχόλιά σας, για τις σκέψεις σας και για το γεγονός ότι ήρθατε εδώ, γιατί άξιζε να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση διότι πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια συνδυασμού στη χώρα σας της σταθερότητας με μεταρρυθμίσεις για να υπερισχύσει ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια, ε, αντίστροφη πορεία και βλέπω ότι και εσείς και ο Βασιλέας προσπαθείτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε τον κόπο να έρθετε να μας επισκεφθείτε. Ευχαριστώ. Well, my friends, we have to continue and we have a... Ας προχωρήσουμε, έχουμε ένα βαρύ πρόγραμμα γιατί πρέπει μέχρι τις 6.30 να τα έχουμε τελειώσει όλα. Πάντοτε είναι δύσκολο να τα βγάλει κανείς πέρα με ε, τις ε, προσωπικότητες τους, τις διάσημες προσωπικότητες. Τώρα λοιπόν έχουμε το, την έκθεση για το Μαυροβούνιο και αν είναι εδώ ο κύριος Τάνο θα τον παρακαλούσα να μας το παρουσιάσει για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει πάρα πολύ φασαρία γιατί ακόμη αδειάζει η αίθουσα. Είναι το δεύτερο ψήφισμά μου και παραμένω στα σχόλιά μου ότι το Μαυροβούνιο παραμένει μία, ένα απλό θέμα και παρακολουθούμε τις ε, εξελίξεις για να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαυροβούνιο ζήτησε το 2008 να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, απελευθερώθηκε το θέμα της ελευθέρας διοικήσεως το 2009 και η χώρα έγινε το 2010 επίσημη υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνεδριάσει όμως απεφασίστηκε να καθυστερήσουν ε, την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων και αυτό οφειλόταν ε, σε πολιτικά κίνητρα και εσωτερικά προβλήματα ορισμένων κρατών μελών και όχι στην πρόοδο του Μαυροβουνίου που είχε προχωρήσει σε 7 βασικούς τομείς ε, και έχοντας δουλέψει σκληρά για να καλύψει τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία άλλωστε το αναγνωρίζει. Οι 7 αυτές τομείς προέβλεπαν ότι έπρεπε να βελτιωθεί η εργασία του Κοινοβουλίου, ε, η ε, επαγγελματική πρόοδος, ανεξαρτησία του, της δικαιοσύνης Κατα καταπολέμηση του εγκλήματος και η κατάρτιση κοινωνίας των πολιτών. Και εγώ αναφέρομαι και στην οικονομία και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει, διότι όσο συνεχίζεται η ε, κρίση της Ευρωζώνης και το Μοντενέγκρο, ε, το Μαυροβούνιο χρησιμοποίησαν νόμισμα το ευρώ χωρίς να είναι μέλος της Ευρωζώνης ε, ε Πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία στη χώρα αυτή για να μπορέσουν να προωθωθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να υπάρξει ανάπτυξη. Ε, έχει, ε, ε, έχει προσχωρήσει σαν πλήρες μέρος στον ΠΟΕ από τον Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους και σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κοιτάξει τις σχέσεις τους και ε, το Μαυροβούνιο είναι μία χώρα με πολύ λιγότερα προβλήματα από ότι ε, οι γειτονές η Κροατία, ε, η Σερβία μετά πριν από 10 χρόνια ανεξαρτητοποιήθηκε και υπάρχει και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης όλα αυτά αναφέρονται ε, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στην ενεργειακή πολιτική και για την δυνητική ε, καταστροφή στο περιβάλλον εάν δημιουργηθεί ένα σιδροελεκτρικό σταθμός με φράγμα και υπάρχει ε, ανησυχία σχετικά με τη διαφάνεια και τις κατηγορίες για διαφθορά στη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεως και πίεση εις τους δημοσιογράφους, άρα αφισβητείται η ελευθερία του τύπου. Είναι όμως ένα παράδειγμα καλής συνεργασίας με τους γειτονές της ε, η χώρα αυτή και ε, έχει λύσει χωρίς ε, ε, προβλήματα το πρόβλημα που είχε για τα σύνορά της που υπευλήθη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει καλές σχέσεις με την Σερβία, την Μακεδονία και την Κροατία. Είναι δηλαδή μια επιτυχής χώρα και Ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2012 όπως έχει ανακοινωθεί. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι οι τέσσερις συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες διαπραγματευτήκαμε χθε καλύπτουν τις περισσότερες από τις 75 τροπολογίες των συναδέλφων που μου φάνηκε ένας υπερβολικά υψηλός αριθμός. Ευχαριστώ. Και τώρα καλό του σκιώδη συγητή τους και συγητές θα μιλήσουν για δύο λεπτά. Παρακαλώ προσπαθήστε να παραμείνετε στα δύο λεπτά. Κύριε Μπρισάτζιτς, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί συμφωνώ με τον κύριο Τάνοκ ότι το Μαυροβούνιο είναι πραγματικά μια ιστορία επιτυχίας και θα ήθελα να τον συγχαρώ και τον κύριο Τάνοκ για το κείμενό του είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο. Ήταν πολύ εύκολο να εργαστούμε ως και ηγητές γιατί επήλθε ευρεία συμφωνία μεταξύ των σκιωδών ε, υποστηρίζουμε όλες τις συμβαστικές ε, τροπολογίες καθώς και την όλη εικόνα που μόλις μας παρουσίασε συγητής. Πολύ καλή δουλειά, συγχαρητήρια και τον ευχαριστώ και εκείνον και τους υπολείπους σκιώδης συγητές για την τόσο καλή συνεργασία και συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φέρμ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα πω και εγώ ότι θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ. Είναι καλή έκθεση, ισορροπημένη, συμβαστικές τροπολογίες, συνεργασία, όπως ε, ακούστηκε για τη διαφθορά, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία των ΜΜΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να κρίνονται με βάση τις δικές σου προσπάθειες και το αποτέλεσμα και η προενταξιακή τους διαδικασία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι προϋπόθεση ή όρος άλλων κρατών. για τη χρηματοδότηση του προενταξιακού μέσου ΙΠΑ η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση και για τις πολιτικές φύλου θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο εκεί. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην κοινωνία των πολιτών, συνδικαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μας ε, υποστηρίζει 100% κύριο Στάνοκ, αλλά η Επιτροπή φαντάζομαι ναι. Εφτά τροπολογίες έχουμε μαζί με τους Πρασίνους και την κυρία Λούνα Τσεκ που θα πει για τα δικαιώματα των LGBT, τα περιβαλλοντικά κτλ. το θέμα είναι είμαστε πολύ αυστηροί ή πολύ επίκης. Νομίζω έχουμε βρει μια καλή ισορροπία. Είναι θετικό το μήνυμα προς το Μαυροβούνιο. Ε, του συγχαίρουμε γιατί έχουν σε μεγάλο βαθμό υλοποιήσει τα κριτήρια ένταξης, αλλά από την άλλη εκφράζουμε τις επικρίσεις και λέγουμε ότι θα πρέπει πολύ περισσότερα να επιτευχθούν σε πολλούς τομείς. Χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες στην υλοποίηση των ε, μεταρρυθμίσεων, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, ε, αυθορά οργανωμένο έγκλημα, αυτά είναι ε, θεμελιώδη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιγκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Τάνοκ, ο οποίος δούλεψε πολύ σκληρά για αυτή την έκθεση. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα θετικό και πολύ ισόρροπο. Εγώ δεν εξεπλάγει με τον αριθμό των τροπολογιών. Ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι συνήθως σε εκθέσεις αυτού του είδους. Πάντως δεν μπορώ παρά να επενέσω τον εισηγητή, διότι συνεργάστηκε στενά μαζί μας, συνδυάζοντας πολλές διαφορετικές ιδέες μεταξύ τους, τις συμβαστικές προτάσεις και δείχνοντας επίοικια τις απόψεις που δεν ήταν κοινέ μεταξύ όλων. Νομίζω εδώ έχουμε μια περίπτωση, μια καλή περίπτωση, θετική, μια της συγκεκριμένη χώρας, η οποία έχει φέρει εις σε αυτά που ανέλαβε. Έχει πετύχει κάποια εσωτερική συνοχή, εθνική συνοχή, ιδίω ω προ την ευρωπαϊκή τη προοπτική. Πρέπει να επενέσω και το ε, Μαυροβούνιο για τη συνεισφορά του στι σχέσει καλή γειτονία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίω πρέπει ακόμη να γίνουν κάποια πράγματα ώστε το νομοθετικό πλαίσιο με νόμους κατά της διαφθοράς, λόγου χάρη, να αρχίσουν να υλοποιούνται. Επίσης κάποια άλλα στοιχεία θα θέλαμε να βελτιωθούν. Όταν μιλάμε για την πίεση εις βάρος των δημοσιογράφων, των εκπροσώπων του τύπου, κάποια περιστατικά που αφορούν εκπροσώπους του τύπου. Εκεί συμφωνώ με άλλους ε, συν εισηγητές και σχεδόν εισηγητές. Το Μαυροβούνιο καλό θα ήταν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις καθώς και την επόδυνη πορεία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ για την εργασία την οποία έκανε για την παρουσίαση του ψηφίσματος, της εκθέσεως μάλλον και ε, για τον τρόπο με τον, οποίο ελήχθηκε για να βρει συμβιβαστικές λύσεις. Καλό θα είναι να διακηρύξουμε ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει το να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση του Μαυροβουνίου πριν από το καλοκαίρι. Και έτσι θα επιληθούν και τα προβλήματα της διαφθοράς και τα λοιπά όταν θα έχουν λυθεί τα προβλήματα του άρθρου 23-24. Σχετικά με αυτά που είπε ο συνάδελφος Φέρμαν, είμαστε πολύ επίκης, ήθελα να σας πω ότι εγώ αυτό το οποίο προτείνω, εκτός από αυτά που είπε ο κύριος Τάνο, είναι ότι το, η συμβιβαστική τροπολογία 2 και 4 δεν είναι αρκετές ισχυρές και ε, δεν νομίζω ότι η πρόοδος ήταν τόσο καλή για να τους ανοίξουμε τις αγκάλες τώρα διότι υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις ε, μεγάλης διαφθοράς υψηλού επίπεδου που πρέπει να ληφθεί υπόψη και ακόμη και μέσα στο κείμενο αναφέρεται το γεγονός αυτό αλλά δεν νομίζω ότι η διατύπωση είναι αρκετά αυστηρή και αυτά που είπαν ο συνάδελφος Κούγκαλ και άλλοι σχετικά με την αγορά το, με το θέμα αυτό δεν είναι αρκετά σαφής. Ε, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, αλλά σήμερα ε, θα ήταν καλό να αναφέρουμε ποιοι ασχολούνται με τον ε, τύπο στην, στο Μαυροβούνιο. Σχετικά με το LCBT ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται ε, μόνο ένας ε, νόμος που να καταργεί τις, τις διαφορές και θα ήταν καλύτερο να ενισχύσουμε την διατύπωση η οποία χρησιμοποιείται. Σωστά κύριε Κατανοκασχολείστε ασχολείστε με το θέμα της οικολογίας και των υδροηλεκτρικών ε, ε, ε, φραγμάτων αλλά όπως είπε ο κύριος Βάγκελ και ο κύριος Κάτσιν θα έλεγα να αναφερθούμε στον ηλεκτρισμό και στα ε, φράγματα. Ε, λυπούμε που δεν δεχτήκατε τις τροπολογίες μας, αλλά θα τις, προ... Ε, θα τις ξαναπροωθήσουμε, διότι υπάρχουν ορισμένα θέματα που θα έπρεπε να περιλάβουμε. Ευχαριστώ. κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε μια καλή έκθεση για το Μαυροβούνιο. Ο κύριος Στάνος συνέβαλε στην ποιότητα αυτής της εκθέσεως και προχωρά αρκετά καλά. Οπότε ελπίζω η πρόοδος να είναι ομαλή και να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις προσχωρήσεως εφέτος. Από την αρχή υπήρξαν σοβαρές προ, προοδεί σχετικά με την εργασία του Κοινοβουλίου, το, την εργασία του εκλογικού σώματος, τη χρηματοδότηση των κομμάτων, αλλά συγχρόνως και στην μεταρρύθμιση του ε, δικαστικού συστήματος και ε, στηρίζουμε ε, την προσχώρηση του Μαυροβουνίου. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τάνοκ που μπόρεσε να ε, οδηγήσει συμφωνία και να διατυπώσει τις συμβιβαστικές τροπολογίες και σχετικά με αυτό το οποίο είπε η κυρία Λούνατσεκ στους συμβιβασμούς πρέπει κανείς να περιλάβει ορισμένες ιδέες και τέλος η συμβιβαστική λύση η οποία χρησιμοποιήθηκε είναι καλή και θα έπρεπε να τη στηρίξουμε. Ευχαριστώ κύριε Μπρισάντζης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να πω απλώς ότι υποστηρίζω έντονα όλες τις συμβαστικές τροπολογίες. Κατά 99% η συμβαστική του κυρίου Κούκαν, η τροπολογία του μάλλον καλύπτεται και ο ίδιος θα την αποσύρει. Αυτό που είπε η κυρία Λούνα Τζακενό δηλαδή. Επίσης, μια μικρή πολιτική ομάδα ε, όπως αυτή που εκπροσωπεί η κυρία Λούνατσεκ δέχτηκε πολύ μεγάλη γενοδορία από πλευράς του κυρίου Τάνοκ και ε, ε, σας καλύπτουν οι τροπολογίες. Αν θεωρείτε ακόμα ότι δεν έχουν καλυφθεί, ας ψηφίσουμε τις τροπολογίες σας και να δούμε τι θα πάρει το αποτέλεσμα. Νομίζω καλό θα ήταν να υποστηρίξετε τους συμβιβασμού γιατί καλύπτουν πάρα πολλά από τα όσα ζητάτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόουτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι ήταν ε, πολύ καλή η προσπάθεια του Μαυροβουνίου να ανταποκριθεί στις βασικές προτεραιότητες. Κάτι που είναι σημαντικό και θα αποτελέσει και παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες είναι ότι οι βασικές πολιτικές δυνάμεις συνεργάζονται στη χώρα αυτή για ένα στρατηγικό στόχο που έχουν. Αυτό θα μπορούσε να εμπνεύσει και να ε, ε, βοηθήσει γειτονικέ χώρες όπως για παράδειγμα την Αλβανία. Ε, το Μαυροβόνιο έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη σταθεροποίηση της οικονομίας του και η μακροοικονομική σταθεροποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική δεδομένης και της σημερινής οικονομικής κατάσταση στην Ευρώπη. Η έκθεση του κυρίου Τάνοκ με ξεκάθαρο τρόπο παρουσιάζει την κατάσταση εκεί και δείχνει ποια είναι τα προβλήματα που παραμένουν στη δικαιοσύνη, στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπάρχουν ακόμα αδυναμίες, αλλά αξίζει να αναφέρουμε και να τονίσουμε ότι το Μαυροβούνιο δεν θα μπει αύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει χρόνο να αλλάξει, να αναπτυχθεί και στο βαθμό που οι βασικές πολιτικές δυνάμεις αφιερώσουν όλοι τους την προσπάθεια στις προτεραιότητες αυτές, είμαι βέβαιος ότι μόλις αρχίσουν οι προενταξιακές διαπραγματεύσεις θα ε, συνεχιστεί η σημαντική πρόοδο. πρόοδο είναι πολύ ευχάριστα αυτά που μαθαίνουμε από το Μαυροβούνιο και επαναλαμβάνω, είναι παράδειγμα προς μίμηση από γειτονικέ χώρες και μεταξύ αυτών σκέφτομαι εδώ και την Αλβανία και τη Βοσνία Ζεγοβίνη και τη Σερβία για την ομοψυχία των πολιτικών δυνάμεων. Συγχαρητήρια λοιπόν και στο Μαυροβούνιο αλλά και στον κύριο Τάνοκ. Κυρία Λούνατζεκ, 30 δεύτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Μπρισάτζης. Έχετε δίκιο. Πολλά ε, είναι εκείνα στα οποία συμφωνεί ο κύριος ε, Τάνο. Και επίσης δεν είμαστε μικρή ομάδα. Εγώ θα μας χαριστεί ε, τη ρίζα μεσαίου μεγέθους πολιτική ομάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια κριτήρια για την ε, ένταξη σε αυτή για να πιέσει τις χώρες να κάνουν πρόοδους. Και αυτό θέλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απαντώ λέγοντας ότι Χαίρομαι που ο κύριος Τάνοξη έλαβε τόσα πολλά από τις προτάσεις μας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επικριτικοί. Εντάξει, ο, ο εισηγητής τώρα για να διευθετήσει αυτό το θέμα. Δεν θα μπω εγώ σε αυτά τα χωράφια αντιπαράθεσης πρασίνων ε, με το ΕΛΚ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πρισάτζης. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια Έχουμε πάει μαζί επανειλημμένα στη χώρα. Είναι πραγματικά εμπειρογνώμων και σέβομαι τη σοφή της άποψη και αντίληψη για τα όσα συμβαίνουν στο Μαυροβούνιο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φέρμ. Συμφωνώ με το σχόλιο σας ότι κάθε χώρα θα πρέπει να κρίνεται από τις ίδιες επιδόσεις και να μην έχουμε γενική κρίση. Βεβαίως, εγώ θέλω να υποστηρίξουμε κάθε είδος μέτρα κατά των διακρίσεων διαφορών μειονοτήτων, γυναίκες, ε, συνδικάτα, LGBT κτλ. Ε, αυτά τα αναφέρω. Και όπου υπάρχει πρόβλημα, ε, θα το δούμε στην εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων. Δεν θέλω όμως να επισκιαστούν όλα τα άλλα από αυτό το στοιχείο στην έκθεσή μου. Είναι ευρύτατη η έκθεση και έχει να κάνει με την πρόοδο της χώρας προς την ένταξη καταπολέμηση της διαφθοράς βεβαίως ε, ε, είναι κάτι που με απασχολεί και εμένα και τους συναδέλφους για τα Δυτικά Βαλκάνια και οι παρενοχλήσεις και οι δολοφονίες φερόμενες των δημοσιογράφων είναι πολύ σοβαρό. Κύριε Λούνατσεκ, αν τη διατύπωση των συμβιβασμών, γιατί λέμε ότι καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε την περαιτέρω πρόοδο στην υιοθεσία ε, στην έγκριση μάλλον της νομοθεσίας κατά το διακρίσιο. Στην έγκριση είμαστε, στην εφαρμογή δεν έχουμε φτάσει. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι υπάρχει τώρα νομική βάση, νομικό πλαίσιο ε, για να συνεχιστούν τα βήματα πρόοδου. Δεν ξέρω, ίσως είναι παρεξήγηση τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο συμβιβασμός. Τώρα, ε, να κατονομάζονται και να διαπομπεύονται εταιρείε. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τις εταιρείε ε, τηλεπικοινωνιών, αλλά δέχομαι ε, επιστολές και για άλλες εταιρείες που θεωρούν ότι ε, ξαπάτησαν ορισμένους ε, επενδυτές και μάλιστα μερικοί από αυτούς ε, διαμένουν στην εκλογική μου περιφέρεια στο Λονδίνο. Αλλά αυτό θέλω να το δω διμερώς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη χώρα και την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου αλλά δεν θέλω να κατονομάσω εταιρείε τώρα στην έκθεσή μου. Το συζήτησα και με την Άννα και με του φιλελευθέρου. Και επίση, επειδή δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία, δεν θα μπούμε τώρα σε μια τέτοια διαδικασία ονοματολογία στην έκθεση. Τώρα για τους υδροελεκτρικούς σταθμούς και τα φράγματα έχω κάποιες επιφυλάξεις αλλά είναι και μια πηγή συναλλάγματος ε, για το Μαυροβούνιο για να μπορεί να εξαγάγει ηλεκτρική ενέργεια και προς την Ιταλία και άλλες χώρες. Δεν μπορώ να αποκλείσω αυτό το μοντέλο ως ανάπτυξη. Ε, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορείτε να κάνετε πράσινη τέτοιες τροπολογίες, αλλά θα τις καταψηφίσω. Κύριε Κούκαν, σας ευχαριστώ. Είστε από τους μεγαλύτερους εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου μας για την περιφέρεια και ό,τι λέτε λαμβάνετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Και τον κύριο Ρότσεκ τώρα έχετε απόλυτος δίκιο. Το έχουμε πει, το Μαυροβούνιο δεν έχει καμία σχέση με τα εσωτερικά προβλήματα που έχουν οι γείτονες. Αναφερθήκατε στην Αλβανία με, με το συνεχιζόμενο διχασμό στο εσωτερικό της χώρας, ε, στο Μαυροβούνιο. Ε, αυτά δεν συμβαίνουν. Όπως είπατε, δεν θα μπουν αύριο στην Ένωση Μαυροβούνιο, ούτε καν έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις. Όταν αρχίζουν να ανοίγουν και να κλείνουν τα κεφάλαια, εκεί θα γίνει πραγματική και σημαντική ε, διαπραγμάτευση και τότε θα έχει έρθει ώρα να δούμε κατά πόσο εφαρμόζονται οι νόμοι που εγκρίνονται. Προς το παρόν χρειάζεται να στηθεί ένα νομικό πλαίσιο και να βοηθήσει και το Κοινοβούλιο και μετά στα επιμέρους κεφάλαια θα δούμε τι ε, ισχύει. Ευχαριστώ όλους σας για τα καλά σας λόγια και την υποστήριξη και προσβλέπω αύριο στην ψηφοφορία και στην έγκριση του ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Tano. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Ωραία. Προχωρούμε αμέσως στο επόμενο θέμα που είναι το σχέδιο έκθεσης συνοδευόμενο από πρόταση σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις λεπτομερείς όρους πιθανής λειτουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία. Πέντε λεπτά, κύριο Λάμπστορφ. Ευχαριστώ. Το κύριε Πρόεδρε. Ε, πρόκειται ε, εδώ για μία κίνηση προς το Συμβούλιο, δηλαδή ε, θέλουμε να δείξουμε ποια είναι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μία κοινοβουλευτική δημοκρατία και κατόπιν των συζητήσεων που είχαμε τους τελευταίους μήνες προσπάθησα όλα αυτά να τα παρουσιάσω όσο το δυνατόν πιο πιο γενικά και ε, να συγκεράσω τα διάφορα ενδιαφέροντα και συμφέροντα διότι στην αρχή είχε ξεκινήσει μία θεωρητική συζήτηση που τώρα έχει μεταβληθεί σε μία συγκεκριμένη κίνηση ε, οι υπηρεσίες προχωρούν θετικά και περιμένουμε να έχουμε ένα καταστατικό κατά τον Ιούνιο και γι' αυτό ε, είναι η κατάλληλη στιγμή να ε, καταρτήσουμε αυτή την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Δημοκρατία. Ε, υπάρχουν τροπολογίες στο αρχικό κείμενο που ήταν επικοδομητικές. Από κοινού έχουμε καταρτήσει ήδη 12 συμβιβαστικές τροπολογίες, έχουν συζητηθεί και κατά 95-96% υπάρχει συμφωνία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι εδώ να τονιστεί η προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, ε, ποιοι είναι οι αποδέκτες ε, των κινήσεων και παροχών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία. Είναι οργανώσεις που μέχρι στιγμή δεν μπορούσαν να στηριχτούν ή που είχαν δυσκολίες να στηριχθούν διότι παραδείγματο χάρη δεν ήταν πρόσωπα νομικού δικαίου, είχαν διοικητικά προβλήματα ή τέλος πάντων άλλα προσκόμματα. Θέλουμε εδώ να τονίσουμε και κάτι παραπάνω πέραν της ευελιξίας που είναι ένα βασικό στοιχείο αυτής της προστιθέμενης αξίας. Ε, ιδίως σε μία μεταβατική περίοδο είναι δύσκολο κάποιοι οργανισμοί να έχουν ε, ε, χρηματική στήριξη και αυτό το Ίδρυμα μπορεί να συμβάλλει και να συνεργαστεί τα πλαίσια αυτά. Γι' αυτό και ε, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε επικαλύψεις με άλλα ισχύοντα συστήματα όπως το Ευρωπαϊκό Μέσον Δημοκρατίας για να έχουμε μία ευέλικτη αποτελεσματική μικρή δομή η οποία ε, ε, θα ιδρεύει στις Βρυξέλλες θα μπορεί να συνεργαστεί και επί τόπου και με πολιτικά ιδρύματα, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ούτω καθεξής. Τρίτο σημείο στο οποίο όλοι συμφωνούμε, όταν χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει ο, ε, ε, ε, δημοσιονομικός κανονισμός να γίνεται πλήρως σεβαστός, σεβαστός και αυτό έχουμε συμφωνήσει όλοι. Επιπλέον το Κοινοβούλιο θα πρέπει και μετά από την κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία Δημοκρατία να συνεχίσει να εμπλέκεται και να υπάρχει μία ισοσκελισμένη εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις δομές του Ιδρύματος αυτούς κατά τρόπο ώστε να μπορέσει να συμβάλλει θετικά και να διαμορφώνει και το πρόγραμμα. Θα πρέπει πέραν αυτού να υπάρχει και πολιτική εποπτεία και να ε, υπάρχει μία παρουσία και Απολογισμός στην Επιτροπή μας κάθε χρόνο. Αυτό που θα ψηφίσουμε αύριο είναι ε, τι ε, μπορούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αδύναμες μικρές νέες δομές και αυτό θα πρέπει να γίνει πολυμερός και είναι σαφές για να στηρίξουμε πολιτικές κινήσεις χωρίς όμως να θεωρήσουμε σαν κριτήριο ότι θα διακόπτεται η ενίσχυση όταν η κίνηση θα μετατρέπεται σε πολιτικό κόμμα. Αλλά όπως σας είπα κατά 95% έχουμε συμφωνήσει όλοι και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία οπότε προσβλέπω αύριο αύριο στην ολοκλήρωση αυτής της καλής εργασίας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε. Κυρία, Κυρία Σαϊφή, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Λάμπστορφ και για την ποιότητα της εκθεσής του και για το πνεύμα συνεργασίας στις συζητήσεις μας. Μπορέσαμε έτσι να συνοσπιστούμε γύρω από ένα τέτοιο σημαντικό εγχείρημα, τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία. Οι πολιτικές ομάδες έχουν καταλήξει κάποιε συμβιβαστικέ λύσει και πέραν ενό ευαίσθητου σημείου που θα σας παρουσιάσω ευθύ αμέσω. το πολύπλοκο αυτό εγχείρημα δεν φαίνεται να σκοντάπτει σε κάποια μείζωνα δυσκολία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό γιατί το Ευρωκοινοβούλιο έχει κατανοήσει την σημασία του όλου θέματο και έχει υπάρξει ιδιαίτερα ταχύ στην αντίδρασή του. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να είμαστε αποτελεσματικοί. Το να δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία σήμερα θα προκοδοτήσουμε την Ένωση με ένα μέσο γρήγορη αντίδραση, ευέλικτο και προσαρμοσμένο στι σημερινέ προκλήσει τη δημοκρατία, δηλαδή τι ε, θεσμικέ και συνταγματικέ μεταρρυθμίσει, τον πολιτικό την πολιτική πολυφωνία και τις ε, εκλογικές προσδοκίες σε πολλές χώρες. Θα ήθελα τώρα να φτάσουμε στο αμφιλεγόμενο σημείο της έκθεσης του κυρίου Λάμστορτ, Ζήτημα του καταλόγου των δικαιούχων του Ιδρύματο. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συζητήσεών μα, ο εισηγητή καθώ και ένα μεγάλο μέρο βουλευτών θύμισαν ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε οικονομικά το σύνολο των ε, φορεών που είναι υπέρ τη δημοκρατία στι ε, χώρε σε δημοκρατική μετάβαση. Εγώ στηρίζω πλήρω την ιδέα αυτή και κατά τα άλλα συνεννοηθήκαμε και κατά το πρώτο τμήμα τη συμβαστική πρόταση 5 ώστε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των δικαιούχων ένας αριθμός φορέων όπως οι δημοκρατικοί ακτιβιστές, οι ε, blogger, οι στατευμένοι καλλιτέχνες και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Για το ευαίσθητο αυτό σημείο, να θυμίσω ότι οι χώρες που θέλουμε να, βοηθήσουν, να βοηθήσουμε ε, έχουν ε, πρέπει να καταστήσουν σεβαστή την αυτοκυριαρχία τους, την αυτοδιάθεσή τους. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς ε, στις πολιτικούς, στα πολιτικά κόμματα των χωρών αυτών να προσφέρουμε στήριξη ακόμα και αν είναι καινούρια ή παλιά. Εδώ έχουμε μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια να κατηγορηθεί για παρεμβολή. Η συμβαστική πρόταση λοιπόν 5 θα ψηφιστεί ξεχωριστά για το κατά πόσον θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να αναφέρονται στον κατάλογο των δικαιούχων ή όχι. Νομίζω ότι αυτή η συμβαστική λύση είναι ένας επιδομητικός ε, τρόπος συμβαστική λύση και η ψηφοφορία τη είναι ένα επιδημοτικό τρόπο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να ολοκληρώσω λέγοντα ότι το ίδρυμα αυτό θα πρέπει να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εξωτερική μα πολιτική, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε και να αποκριθούμε άμεσα με συγκεκριμένε αρμοδιότητε. Σα ευχαριστούμε, κυρία Γκόμε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που φτάσαμε ήδη σε αυτό το στάδιο της όλης συζήτησης για αυτή την πρόταση, γιατί νομίζω ότι ήμουν η πρώτη που είχα υποβάλει ε, είχα προβάλει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία από την έκθεση Χάουι του 2010. Να πω λοιπόν ότι τώρα ομιλώ εκ μέρους της ομάδας μου, όχι μόνο ε, για την προσωπική μου άποψη και βεβαίω εκ μέρου τη κυρία Ντεκάιζερ, η οποία ήταν εδώ σήμερα και έχει εργαστεί ω κοιόδηση συγκήτρια για το θέμα αυτό και εγώ και εκείνη θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον κύριο Λάμστροφ για το εξαιρετικό του έργο. Βεβαίω το ίδιο και για τους σχεδόντες εισηγητές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Υπάρχει ευρεία συμφωνία όπως ε, αναφέρθηκε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα ίσονος που έχουν όμως ακόμα τη σημασία τους για την ομάδα μου το πλέον σημαντικό είναι το κατά πόσον θα υπάρχουν δωρεές σε πολιτικά ε, θεμέλια ε, Θα πρέπει αυτό βεβαίω ε, να το αποσαφηνίσουμε με του συζητητέ και του σκιώδει συζητητέ. Επίση, είναι νομίζω καλή η λύση που βρέθηκε για την πολιτική ισορροπία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό για μας ήταν πολύ σημαντικό θέμα και για το ζήτημα των πολιτικών κομμάτων. Εδώ μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις η δική μας όδηση συγκεντρία, η Βερονίκ, θεωρεί ότι λίγο πολύ βάσει των όσων είπε και η κυρία Σέιφη, προτιμότερο θα ήταν να μην προβλέπονται δωρεέ ε, άμεσε τουλάχιστον προ τα πολιτικά κόμματα, αλλά σε φορεί, ακτιβιστέ, προτού προσχωρήσουν σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Πρέπει να πω προσωπικώ, πιστεύω, ότι προκειμένου να διατηρηθεί πολιτική ισορροπία στο Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό να βρούμε εδώ μια λύση. Φανταστείτε να συμφωνούσαμε όλοι. Φανταστείτε, φανταστείτε μια κατάσταση σαν την Νότια Αφρική πριν το τέλο του Απαρτχάιντ. Προφανώ και ήταν σημαντικό τότε να χρηματοδοτηθεί η κίνηση για την απελευθέρωση από το Απαρτχάιντ. Αλλά κάτι ανάλογο θα πρέπει να γίνει και με τη λύση που θα βρεθεί για τη συμμετοχή των γυναικών, καθώ και τον δημοσιονομικό έλεγχο που θα μπορεί να ασκεί το Κοινοβούλιο καθώς και την απονομή των δωρεών με διαβουλεύσεις, μετά από διαβουλεύσεις με αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, Διευθύνουσα Επιτροπή του Ιδρύματος. Αυτό ακόμη πρέπει να ε, αποσαφενιστεί, αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει πολιτική ισορροπία. Ευχαριστούμε, κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ παραμένω στην αρχική μου αξιολόγηση ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία δεν με ικανοποιεί καθόλου, το κατακρίνω και απορρίπτω τελείως ένα τέτοιο οικοδόμημα διότι δεν συνάδει με το δημόσιο το διεθνές δίκαιο και επιπλέον το, το σχέδιο αυτό υποθάλπει το δικαίωμα της κυριαρχίας. Ε, νομίζω ότι είναι κάτι μονοπλευρό το οποίο προωθείται από πολιτικά κόμματα και ε, δείχνει, αποκαλύπτει ποιες είναι οι προθέσεις των υποστηρικτών της κινήσεως αυτής. Γι' αυτό και έχω κάνει μία ριζική η τροπολογία ότι δεν πρέπει ε, να ε, δημιουργηθεί αυτό το ίδρυμα. Επιπλέον η ανεξάρτητη, ε, δεν υπάρχει ανεξάρτητος δημοκρατικός και διάφανος έλεγχος και στηρίζω την συμβιβαστική 10 η οποία λέει ότι όλα τα ιδρύματα αυτού του είδους θα πρέπει να αξιολογούνται από έναν ανεξάρτητο ανεξάρτητο οργανισμό. Πέραν των όσων είπα δεν θέλω να αποφύγω μία επικοδομητική συνεργασία γι' αυτό και έχω προβεί και σε ορισμένες άλλες τεχνικές τροπολογίες τις οποίες έχω υποβάλει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με την εργασία θέλω να ευχαριστήσω τον συντάκτη κύριο Λάμσδορφ ο οποίος προχώρησε με πολύ καλή θέληση και δεν, δεν θέλω μία αντιπαράθεση με την κυρία Λέζιγκ... η οποία εδώ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μία ορολογία του παρελθόντος. Όταν υπάρχει δημοκρατία δεν υπάρχει ε, ε, μία αποκλειστική κυριαρχία των κρατών. Ως εκ τούτου δεν θέλω να εμπλακώ σε μία τέτοια συζήτηση και θα μου επιτρέψετε ε, κυρία Λέζινγκ, να σας πω ότι εγώ δεν αισθάνομαι ότι με αντιπροσωπεύουν τέτοια σχόλια. Θέλω όμως να κάνω ορισμένα ερωτήματα στον κύριο Φων Λάμπστορκ. Πώς θα εξασφαλίσουμε ε, την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδίω όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου. Δεύτερον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε να αποφευθούν επικαλύψεις με άλλα μέτρα, μέσα και άλλα τέτοια ιδρύματα κατά τρόπον ώστε να μην ε, πολλαπλασιάσουμε τη γραφειοκρατία διότι αυτό φοβάμαι ότι στο τέλος θα υπάρξει μία αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων αυτού του είδους. Επίσης ε, κύριε Φον μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ πόσο θα χρηματοδοτηθεί αυτό το ίδρυμα, ποιος ε, θα συμβάλλει με ποιους πόρους και όσον αφορά την εκτελεστική επιτροπή η οποία θα πρέπει να καταρτιστεί και να έχει συγκεκριμένη μορφή πώς ε, θα μπορέσει ε, αυτή η Επιτροπή να συνεργαστεί επικοδομητικά. Στο σημείο 8-6 λέγεται ότι άπαξ του έτους θα συνέρχεται αυτή η Επιτροπή ε, με άλλα, άλλους οργανισμούς και θεωρώ ότι είναι ανεπαρκέστατη αυτή η πρόβλεψη και χρειάζεται να γίνουν πολλά παραπάνω και ενδεχομένως οι τροπολογίες οι οποίες θα ψηφίσουμε αύριο θα επιτρέψουν να ε, ε, συγκεκριμενοποιήσουμε αυτά τα θέματα αλλά ήθελα να σας πω ότι αύριο με την ψηφοφορία θα ξεκινήσει η δουλειά και θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε για να μην παραγωνιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ ο κύριος Τζιπ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το ε, Γκόμι Λάμσοφ για την τόσο ενδιαφέρουσα όσο και καλό διατυπωμένη έκθεση την οποία αύριο καλούμαστε να εγκρίνουμε. Θα ήθελα συγκεκριμένα να τονίσω ότι η Πολωνία πρωτοστάτησε στην πρόταση αυτή ήδη από τις παραμονές της ε, Προεδρίας της. Ήταν εμβληματική πρωτοβουλία και της Πολωνικής Προεδρίας και ερχόταν να απαντήσει σε μια δυναμία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά σε χώρες ε, σε μετάβαση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μετάβαση, όπως το είχαμε δει και σε προηγούμενη έκθεση της κυρίας Δεκεζέρ. Θα πρέπει να υποφεληθούμε από την εμπειρία χωρών που γνώρισαν αυτή τη μετάβαση. Χρειάζεται μια προσέγγιση ευέλικτη. Να ξέρουμε όμως και τι σημαίνει αυτή η ευελιξία. Υπάρχει το Αμερικανικό Ίδρυμα ε, για τη Δημοκρατία που κατάφερε να ε, κρατήσει στη ζωή την αλληλεγγύη στην Πολωνία. Αν δεν υπήρχε αυτή η υποστήριξη το 81 η Solidarnosc δεν θα μπορούσε καν να υπάρξει. Βεβαίως τα κόμματα αυτά ε, δεν είναι κόμματα και δεν μπορούν να εγγραφούν ε, επίσημα γιατί δεν είναι τμήμα του πολιτικού συστήματος μιας χώρας κάποια στιγμή. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε δημοκρατικούς κανόνες εξορισμού, ε, οι χώρες αυτές δεν έχουν πολιτικά κόμματα. Είναι κάποια κινήματα στα σπάργανα, το γεννάστε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολιτικές επιφυλάξεις. Ας πούμε, ε, το καθεστώς του Λουκασένκο στη Λευκορωσία δεν θα χαιρότανε να υποστηρίζουμε εμείς τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Αυτό είναι προφανές, έτσι δεν είναι. Μίλησε κάποιος ε, ε, εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης για κόμματα, νόμιμα, παράνομα, ανθρώπινα δικαιώματα. Και πάρα πολύ γρήγορα καταλάβαμε τι τύχη έχουν οι ηγέτε τη αντιπολίτευση και οι ακτιβιστές που καταλήγουν στη φυλακή. Εμείς θα πρέπει να υποστηρίζουμε τον εκδημοκρατισμό και γνωρίζουμε ότι τα μέσα που έχει στη διάθεσή του το σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ευέλικτα και δεν προσφέρονται για ταχεία απόκριση σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν βοηθούν ε, την αντιπολίτευση. Ευχαριστώ, Κόμις Λάμστορφ, για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι χαίρομαι για την ευρεία υποστήριξη που ακούστηκε από τους συναδέλφους και όδης ή εκπροσώπους, γιατί ορισμένοι κολλείονται, η Βερονίκα προκειμένου, Δεκεζέρ. προκειμενου Κεζέρ, ένα σημείο στο οποίο διαφωνούμε, θα το δούμε στην ψηφοφορία, θα το λύσουμε και θα έχουμε ένα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Στα πιο έτσι, κρίσιμα σημεία να πέρασω στα γερμανικά, γιατί ήταν ο κύριος Πέτερινγκ και η κυρία Λέζινγκ. Ε, κύριε Πέτερινγκ, δεν σας βάζω στο ίδιο τσουβάλι, μην ανησυχείτε. Μακριά από μένα αυτή η ιδέα, δεν θα άρεσε ούτε στην κυρία Λέζινγκ, οπότε είστε ικανοποιημένοι και οι δύο. Ε, για να είμαι και ασφαλής εγώ και όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά. Κυρία Λόζινγκ, είπατε ότι η ομάδα σας έχει βασικές επιφυλάξει, το έχετε ξαναπεί, δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει. Και στι ε, συνεργασίε συμμετείχατε και με τους βοηθούς σα. Ε, ο κύριος Πέτερινγκ έχει την τελευταία εκδοχή του κανονισμού, του καθεστώτος ε, και η έγκριση από ανεξάρτητη τρίτη αρχή είναι δεδομένη. Λοιπόν, κύριε Πέτερινγκ πώς εξασφαλίζονται τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα κάνουμε τη σύσταση. Αν δεν έλεγα κοιτάξτε κάτι τρέχει και πρέπει να κάνουμε εμεί σύσταση, δεν θα γινόταν τίποτα και δεν θα το είχε κανεί και δεν θα είχε πάρει είδηση. Μετά, εκπροσωπούμαστε στην ομάδα εργασία. Ε, με παρακάλεσε ο Έλμαρ Μπρόκ να εκπροσωπήσω εκεί την επιτροπή μα, πράγμα που πράττω. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, τα είπα και εκεί στην ομάδα εργασίας ήδη από την πρώτη συνάντηση. Βεβαίως είναι ο, δημοσιονομικός κανονισμός για ε, τα κοινοτικά μέσα πλήρως και σε ό,τι αφορά την εγγραφή στον προπολογισμό αλλά και την εκτέλεση και τον έλεγχο. Αυτό διαφυλάσσεται και είναι τελείως αναμφισβήτητο. Πώς αποφεύγουμε τις επικαλύψεις. Ε, αυτό είναι το θέμα. Πώς ορίζεται το σημείο συνάντηση του Ευρωπαϊκού ε, Ιδρύματος ε, για τη δημοκρατία. Το είπε και η κυρία Σαϊφή με το ε, ε, EIDHR. Μα εμείς θα πρέπει να υποστηρίζουμε κάποιους φορείς και στη συνέχεια ενδεχομένως να μεταβιβάζεται αυτό. Και αυτό έχει να κάνει και με τη συνεργασία. Θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεωτικά να συναντάτε άπαξ ετησίως και θα πρέπει να το γράφει και το καταστατικό. Αλλά σε ένα καταστατικό δεν μπορούμε να γράφουμε όλες τις περιφερειακές συναντήσεις. Το θέμα είναι να είναι ε, στην, ε, στις Βρυξέλλες να λαμβάνονται ανεξάρτητες αποφάσεις Αυτό αφορά και τις επικαλύψεις με το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, ποιος και πόσα. Το θέμα είναι τώρα η εκκίνηση. Ο κύριος Φούλε από το μέσο γειτονία συμφώνησε να δοθεί η πρώτη μαγιά. Η πολωνική δημοκρατία επίσης έχει δεσμευτεί. Τώρα για το μέγεθος δεν το ξέρω το ποσό. Είναι από 3 μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ και άλλα κράτη-μέλη προσεχώς θα αποφαθούν. Προς το παρόν φτιάχνουμε το καταστατικό, τις συνεισφορές οικονομικέ οικονομικές θα τις δούμε. Θα είναι μεικτή χρηματοδότηση όμως από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση οι συνάδελφοι των Πρασίνων που αποχώρησαν δυστυχώς και ο Έλμαρ Μπρόκ πρότισαν να σκεφτούμε ένα trust fund, ένα ταμείο που να συμμετέχουν και τρίτες χώρες, η Νορβηγία ή η Ελβετία προκειμένου αν το επιθυμούν ή μεγάλα ιδρύματα. Αυτό να το κοιτάξουμε, να το εξετάσουμε. Και ένα τελευταίο, ένα Γκόμες νομίζω το είπε. Απάντηση στη ερώτηση του αδέρφου Ζιπ. Υποστήριξη δημοκρατικών κινημάτων όταν δυσκολεύουν τα πράγματα ας πούμε στο Αφρικανικό Κογκρέσο στην Νότια Αφρική στον αγώνα κατά το Απαρτχάιτ δεν θα έχει κανείς πρόβλημα να τους βοηθήσει. Αλλά το λέει και το καταστατικό και θα πρέπει να το προσέξουμε. Υποστηρίζουμε μόνο φορείς ε, που αγωνίζονται ειρηνικά, χωρίς βία, για τη δημοκρατία. Ε, ε, είναι δημοκρατική και φιλιρινική σκοπή. Βεβαίω δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση τα χρήματα να διαχειριστούν για άλλου σκοπού. Σα ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σα. Ε, προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία. Έχει δίκιο ο κύριο Πέτερινγκ. Από την έγκριση τώρα και μετά δεν τελειώνει. Η δουλειά συνεχίζεται φυσικά και σα ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πρόεδρο. Πρέπει να σα ενημερώσω ότι η κυρία Βερονίκ Ντακεζέρ έστειλε μια τροποποίηση στη προφορική τροπολογία στη συμβιβαστική υπαριθμών 7. Εάν θέλετε παρακαλώ να το κοιτάξετε. Συμβιβαστική 7 προφορική τροπολογία θα σας αποσταλεί έτσι και αλλιώς από τη γραμματεία, αλλά σας παρακαλώ να το κοιτάξετε για να το γνωρίζετε πριν την ψηφοφορία. Και η τελευταία φράση λέγει Ε, επανακατανομή που θα πρέπει να σέβεται και αλλάζει η πολιτική ισορροπία και γίνεται πολιτική πολυφωνία. το political balance γίνεται political plurality. Αυτά ζητάει η κυρία Ντεκεζέ. Και θα σας τα διαβάσει η γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, προχωρούμε αμέσω στην επόμενη έκθεση που είναι του κυρίου Ογκουρεάνου σύναψη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση του φακέλου επιβατό PNR στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Thank you, Chairman. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, οπότε θα προσπαθήσω να απλουστεύσω τα πράγματα. Να ξεκινήσω με έναν χρήσιμο διαχωρισμό. Αυτό που όντως συζητάμε και αυτό που δεν ε, Είμαστε... Δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε σε σχέση με την γνωμοδότηση αυτή. Θα έπρεπε να συζητήσουμε δηλαδή την θέση της Επιτροπής μας για τη συμφωνία αυτή από μια ε, σκοπιά διατλαντική από τη σκοπιά της διατλαντικής εταιρική μας σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των, αναγκαν... των αναγκών μας για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε είναι αν μας αρέσει ή όχι η αμερικανική προσέγγιση του θέματος. Νομίζω πρέπει να αναφέρω σαφώς ότι αυτή η νέα συμφωνία για την οποία απαιτήθηκε ένας χρόνος διαπραγματεύσεων είναι μια σαφής βελτίωση της προηγούμενης, των προηγούμενων εκδοχών της. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης, θα αναφέρω ορισμένα. Τώρα τα, υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στα δεδομένα και διορθωσή του από, τους, από τα άτομα. Μπορεί να, να ασκηθούν και ένδικε ε, διαδικασίες για αποκατάσταση. Επίσης υπάρχει μέθοδος PUS για την ε, μεταφορά των στοιχείων. Η διατήρηση των ε, στοιχείων PNR περιορίζεται χρονικά και υπάρχει ο κανόνα του απορρίτου. Βεβαίω κάποιε από τι δικέ μα προτάσει ήταν πιο φιλόδοξε. Όμω νομίζω συνολικά τα αποτελέσματα πετυχαίνουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέλο, νομίζω ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε το εξή. Ποιε θα ήταν εναλλακτικέ λύσει τι θα γινόταν αν δεν εγκρινόταν αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι χωρίς τη συμφωνία αυτή, κατά πρώτον οι αεροπορικές μας γραμμές θα βρίσκονταν σε μια κατάσταση πλήρους ασάφειας. Θα έπρεπε ακόμη να συμμορφώνονται με τις απαιτήσει PNR των ΗΠΑ, αλλά δεν θα είχαν ένα σαφές πλαίσιο που να τους το επιτρέπουν αυτό. Έπειτα, Οπωσδήποτε δεν θα υπήρχε ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ανταλλαγή στοιχείων PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν και πάλι να, να συνάψουν διμερείς συμφωνίες με μονομένα κράτη-μέλη, πράγμα που θα σήμαινε ότι οι διμερείς αυτές συμφωνίες δεν θα ήταν αντικείμενο εξέτασης από δικής μας πλευράς. Συμπερασματικά λοιπόν από η συμφωνία αυτή καλό θα ήταν να εγκριθεί από όλους μας. Υπάρχουν τέσσερις τροπολογίες. Λίγο πολύ στις γραμμές της συγκατάθεσης ή της άρνησης της συμφωνίας. Εδώ δεν έχω αρνητικές ενδείξεις από την Επιτροπή μας. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση, όχι απόλυτη βέβαια. Δεν υπάρχει φυσικά ομοφωνία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η τάση να υποστηριχθεί η συμφωνία αυτή. κυρία Γκόμες, τώρα, για ένα μισή λεπτό. <laughs> Πρόεδρε, Οπωσδήποτε, κάθε χώρα συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ μπορεί να καθορίζει του όρου ε, βάσει των οποίων θα δέχεται πολίτε άλλων χωρών στο έδαφο τη. Έχουμε όμω και άλλο ένα προηγούμενο, το νομικό προηγούμενο, τη συμφωνία PNR με την Αυστραλία. Παρ' όλα αυτά, το προηγούμενο αυτό δεν είναι κάτι που οδήγησε στο θέμα που τώρα εξετάζουμε. Δεν υπάρχει Καμία, καμιά μορφή διαπραγματεύσεων που να είναι τέλειε, ιδίω αυτέ οι τωρινέ, σε σχέση με τι διαπραγματεύσει που είχαμε με την Αυστραλία για την προστασία των δεδομένων των πολιτών μα. Αυτό ήθελα να το σχολιάσω, είτε αυτή την εβδομάδα είτε την προηγούμενη. Το έχω ξεχάσει στην με την παρουσία τη Επιτρόπου Μάλστρομ στην ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Αλλά η καθήλυνα αρμόδια εισηγήτρια, η κυρία Ινφελτ, ζήτησε εξηγήσει για τα πρότυπα ε, των ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών μα και εξήγησε γιατί θεωρεί ότι δεν καλύπτονται πλήρω. Κατά τα άλλα, όμω, θα συμφωνήσω με τον εισηγητή μα, ο οποίο σωστά επισημαίνει ότι η εναλλακτική είναι σαφώ χειρότερη. Θα καταλήξει σε διμερεί συμφωνίε που έχουν διαπραγματευτεί με εθνικέ κυβερνήσει ΗΠΑ που είναι πραγματικά χειρότερε ω προ την προστασία δεδομένων των πολιτών μα. Και προφανώ είναι αδιανόητο να σταματήσουν να πετούν τα αεροπλάνα. Άρα ήταν κάτι που θα έπρεπε να το περιμένουμε. Εγώ ανησυχώ προσωπικά για κάτι που ανακάλυψα ότι δεν βρίσκει σύμφωνε στι ΗΠΑ. Δηλαδή, ενώ τη συμφωνία θα πρέπει να την, κυρώσει, να την εγκρίνει το κοινοβούλιο μας, και ενώ έχουν εγκριθεί συμφωνίε από εθνικά κοινοβούλια διμερό, στην περίπτωση αυτή για τι ΗΠΑ εδώ έχουμε απλώ μια διοικητική συμφωνία, όπω την ονομάζουν εντό εισαγωγικών. Δηλαδή το Κογκρέσο δεν εμπλέκεται. Άρα, εάν αν το επιτρέψουμε, γιατί θεωρούμε ότι οι εναλλακτικέ λύσει είναι χειρότερε για του πολίτε μα, οπωσδήποτε θα πρέπει προηγουμένω να βεβαιωθούμε ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στην όλη διαδικασία αναθεώρηση, η οποία είναι ζωτική σημασία. Θα πρέπει να πιέσουμε. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να διορθωθούν όσα έχουν πάει άσχημα. Πρόεδρος κύριος Νταφ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω ότι ότι η συμφωνία την οποία έχουμε μπροστά μας είναι μια σχετική βελτίωση της προηγούμενης εκδοχής της, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο αυτή που έχουμε με την Αυστραλία και σίγουρα ε, έχει πολλές ε, ελλείψεις. Πρώτα απ' όλα το πεδίο της συμφωνίας. Είναι ιδιαίτερα σαφές. Και στο άρθρο 4.4 θα επιτρέπεται τα στοιχεία PNR να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει δικαίωμα ε, άσκηση ελέγχου στην όλη διαδικασία. Από νομική πλευρά. δεν είναι το σύστημα ασφαλισμένο ούτε συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Θεωρώ ότι δεν ε, βελτιώνονται έτσι οι διατλαντικές σχέσεις και μάλιστα θα αποτελέσει και ένα προηγούμενο αρνητικό για μελλοντικές συμφωνίες PNR με άλλες ενδεχομένως τρίτες χώρες. Χώρες που μπορεί να έχουν ε, κατώτερα συστήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων από τις Ηνωμένες Το να μην αποδεχθούμε τη συμφωνία ίσως ενισχύσει το μελλοντικό ρόλο και την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής στη συμμετοχή της σε περαιτέρω διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Όμως, επειδή η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε τα πολύ αυστηρά πρότυπα που είχε θέσει στο Κοινοβούλιο και στις προσδοκίες του, αυτά που τη ζητήσαμε δηλαδή να πετύχουν, Υπάρχουν και όλες αυτές οι τροπολογίε ε, εκ των οποίων αυτές προτείνουν να απόσχουμε από τη Συμφωνία PNR. Κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ. δεν νομίζω ότι αυτή θα είναι η πρώτη συμφωνία η οποία θα σέβεται τις προδιαγραφές του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι μία από τις συμφωνίες όπου δεν γίνονται σεβαστές οι προδιαγραφές του Κοινοβουλίου και ε, είναι μία βελτίωση όμως ε, σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε στο παρελθόν. Μικρή μεν βελτίωση αλλά πάντως είναι μία βελτίωση. Αυτό το οποίο θα χρειαστούμε είναι να υπάρξει μία απάντηση σε ένα ερώτημα το οποίο δεν είχαμε απαντήσει στο παρελθόν. Μέχρι ποιου σημείου θέλουμε να προασπίσουμε την ασφάλεια και μέχρι ποιου σημείου θέλουμε να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν νομίζω ότι είναι ισοσκελισμένο το κείμενο αυτό σε αυτή την άποψη και αυτό δυσκολεύει την εφαρμογή της συμφωνίας διότι οι συμφωνίες για την αποθήκευση των δεδομένων, οι κανόνες που θα διέπουν αυτές τις ρυθμίσεις, ο χρόνος που θα παραμείνουν και ε, ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν που δεν θα σέβεται τις, ε, τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει είναι κάτι το οποίο ε, επιζητείται για να βελτιωθεί η ασφάλεια λέγεται. Πιστεύουμε όμως ότι ο καθένας μόνος του θα πρέπει να μπορέσει να αποφασίσει κατά συνείδηση. Και εγώ είμαι υπέρ της συμφωνίας διότι αποτελεί ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ ε, μιλάμε ε, για ένα θέμα πολύ λεπτό διότι ε, ξέραμε, ξέρουμε τι έγινε με το SWIFT, βλέπουμε τι γίνεται με το ACTA και βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά με διάφορους συμβαλόμενους ε, ε, μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εισηγητής λοιπόν μας λέει το εξής, ότι η περίοδος ε, κατά την οποία θα διατηρηθούν τα στοιχεία αυτά έχει μειωθεί. Το ερώτημα είναι μέχρι ποιου σημείου. και πώς συγκρίνεται αυτό εάν το συγκρίνουμε με τη συμφωνία με την Αυστραλία. Είναι κρίσιμο σημείο και πολύ σωστά είπε ο κύριος Ντάφ ότι τα στοιχεία τα οποία διατηρούνται μπορούν να μεταδοθούν και αν μεταδοθούν σε ποιον θα μεταδοθούν. Και δεύτερον, άπαξ και μεταδοθούν τα στοιχεία αυτά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που είναι ευαίσθητος με το οποίο δεν ε, συμφωνούμε. Αυτό θα πρέπει να ε, υποβληθεί στον διαμεσολαβητή. Ενδεχομένως η μεταφορά των στοιχείων να μην δημιουργήσει πρόβλημα αλλά ενδεχομένως να ε, παραβιάζει σημαντικά τα δικαιώματα των, των πολιτών και αυτό είναι που με απασχολεί εμένα. Ο κύριος Ουγγουράνου. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα, διότι ε, νομίζω βέβαια αντιλαμβάνουμε αυτές τις ανησυχίες νομίζω ότι ε, επιδέχεται βελτίωσης ε, βελτιώσεις αυτή η συμφωνία πάντοτε όμως θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις και θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις για να απαντήσω στον κύριο Γκάλνις όσον αφορά το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ας απαντήσουν αυτοί για τα δικά τους. Αλλά προς τον κύριο επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν τέλειες διατάξεις για κανένα θέμα και ιδίως σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να συγκρίνουμε με τη συμφωνία με την Αυστραλία διότι δεν μπορούμε ε, να συγκρίνουμε το ποσοστό κινδύνου ε, της Αυστραλίας με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, και όσον αφορά την ε, διαμάχη μεταξύ της ασφαλείας και της ιδιωτικής ζωής, πρέπει να πω ότι είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μία βελτίωση. Μας ζητήσανε να έχουμε μία συγκεκριμένη ε, διάρκεια διατηρήσεως των στοιχείων ε, και αντιλαμβάνομαι ότι ε, θα περιορίζεται μετά από ένα εξάμεινο βαθμιαία η πρόσβαση στα στοιχεία μπορούν όμως να διατηρηθούν σε περίπτωση διεθνών εγκλημάτων μέχρι 10 ετών και τρομοκρατίας μέχρι 15 ετών και εφόσον πρόκειται ε, για ιδιωτικά χεία αυτά θα καταστρέφονται. Σας ευχαριστώ. Και τώρα περνούμε στο επόμενο θέμα. Είναι η εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρέχουσα πρακτική και μελλοντικές προοπτικές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Θα παρακαλώ τον κύριο Σαλαβράκο, συντάκτη γνωμοδότηση, να κάνει μια εισαγωγή. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφους και σκιώδεις ηγητές για τη συνεισφορά τους μέσω της κατάθεσης τροπολογιών αλλά και της επικοδομητικής συνεργασίας για τη σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών. Οι περισσότερες τροπολογίες οι οποίες υπευλήθησαν έγιναν δεκτές καθώς θεωρώ ότι βελτιώνουν το κείμενο και το καθαρούν το καθιστούν πληρέστερο. Η μακροπεριφέρεια της Βαλτικής θάλασσας, η οποία δρομολογήθηκε το 2009, ενέπνευσε και άλλα σχέδια, ένα από αυτά είναι η μακροπεριφέρεια του Δούναβη, που απετέλεσε ένα πρώτο βήμα προόδου, ενώ προβλέπονται και άλλες μακροπεριφέρειες. Σε γενικέ γραμμέ θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκέ μακροπεριφέρειε είναι σημαντικέ για την επίτευξη ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία στα ευρωπαϊκά έργα και συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενός περιορισμένου αριθμού εμβληματικών πρωτοβουλειών συμπληρωματικά με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Με την παρούσα γνωμοδότηση εκφράζεται η γνώμη της Επιτροπής για την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης, τις πρακτικές και τις προκλήσεις κυρίως στη Μεσόγειο θάλασσα. Μερικοί τομεί συνεργασία για τη νέα μακροπεριφέρεια θα μπορούσαν να είναι τα δίκτυα ενέργεια, η επιστημονική συνεργασία και καινοτομία, ο πολιτισμό, η εκπαίδευση και κατάρτιση, ο τουρισμό το εμπόριο, η προστασία του περιβάλλοντο, οι βιώσιμε θαλάσσιες μεταφορέ, η θαλάσσια ασφάλεια και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντο από τη ρήπανση, την υπεραλίευση και την παράνομη αλία. Κάθε μακροπεριφερειακή στρατηγική έχει διπλή διάσταση μια εδαφική λόγω του προσδιορισμού ενός κατάλληλου εδαφικού πλαισίου εφαρμογή και μια λειτουργική μέσω του καθορισμού των προτεραιοτήτων. Πρέπει και οι δύο στόχοι να επιτυγχάνονται για να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η επιτυχία της μακροπεριφέρειας. Έγινε προσπάθεια μέσω των συμβαστικών τροπολογιών να καταστεί σαφές ότι η ακριβής οριοθέτηση της νέας μακροπεριφέρειας ή των νέων μακροπεριφερειακών περιοχή της Μεσογείου δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας γνωμοδότησης καθώς κάτι τέτοιο ε, θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαβούλευσης μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών φορέων, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και τις αρχές της καλής συνεργασίας. Είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω τις απόψεις και των συναδέλφων και των εισηγητών τους οποίους και ευχαρίστησα. Τονίζω ιδιαίτερος ότι υπάρχει μια δέσμευση στο θέμα του χειρισμού των μακροπεριφερειών, ότι οι μακροπεριφέρειες στηρίζονται στο τρίπτυχο όχι νέοι θεσμοί, όχι νέα νομοθεσία, όχι νέοι πόροι και επομένως δεν μπορεί να ε, επαυξήσουμε ε, τη δράση την οποία πρέπει να προβλέψουμε διότι οι μακροπεριφέρειες πιστεύω ε, σε τελική ανάλυση θα αποτελέσουν ε, μελλοντικά μια καλή λειτουργία των της Περιφέρειας της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα είναι γνωμοδότηση. Επί της ουσίας στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή. Θέλουν συνάδελφοι το λόγο να πούν τίποτα. Ναι. Παρακαλώ κύριε Λόπε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαβράκο που δέχτηκε τις τροπολογίες μας, τροπολογίες που καταθέσαμε εμείς σοσιαλιστές, ορισμένα μέλη για να επεκταθούν οι μακροπεριφέρειες όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στη Δυτική. Γιατί έχουμε κοινή ιστορία, κοινή παράδοση, κοινή γεωγραφία, κληρονομιά και η μακροπεριφέρεια είναι πολύ πιο ε, στιβαρή αν περιλαμβάνει και εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Είναι πάρα πολλά τα κοινά θέματα, θα τα δούμε και στο μέλλον. Μερικά πρόσφατα μας έφεραν πιο κοντά, ας πούμε η γεωργική συμφωνία με το Μαρόκο, αλλά και άλλα θέματα μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά και η κοινή μας θέση είναι σημαντική για να μπορέσουν να κινητοποιηθούν έργα και σχέδια που μπορεί ήδη να έχουν κάποιο προπολογισμό, αλλά είναι πολύ σημαντική η συνεργασία και η συνέργεια, όπως λέμε. Σας ευχαριστώ ρητά πραγματικά, κύριε Σαλαβράκο, που δεχτήκατε τις απολογίες μας και επίσης ευχαριστώ όλους όσοι συνεισέφεραν με τροπολογίες στον εμπλουτισμό του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να απαντήσετε, φαντάζομαι. Θέλετε. Πώς ανταποδίδω τις ευχαριστίες μου στη συνάδελφο. Okay, Καλά, σου ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε. Ενημέρωση από τον κύριο Σαλαφράγκα για την αντιπροσωπεία του Χόξ στη Λιβύη το, το Φεβρουάριο. Ναι, αλλά πρώτα είναι ο κύριος Λάμστροφ. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Σαλαφρανκά, έχουμε τον κύριο Λάμστροφ προηγουμένω για τη Νέα Υόρκη και μετά εσείς. Εγώ φταίω, έκανα λάθο, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριο Λάμστροφ. Συγγνώμη Νάτσο, <laughs> θα τα πει μετά. Ήθελα να σας πω σύντομα για την αντιπροσωπεία που πήγαμε ε, στη Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη, τρεις τομείς, γεωγραφικός, θεματικός και θεσμικός, ε, Παλαιστίνη, Αραβική Άνοιξη και η Δυτική Σαχάρα ήταν τα γεωγραφικά, θεματικά ε, ε, η ευθύνη για προστασία και η πολιτική ε, των ΗΕ για την υποστήριξη της δημοκρατίας και τα θεσμικά, τα εσωτερικά των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Το Νοέμβριο πήγαμε, ήταν η κοινή αποστολή, πρέπει να σας πω, πολύ ωραία, με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, είχαμε και ξεχωριστή ενημέρωση για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με το τελευταίο. Το καθεστώς της Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, όταν πήγαμε εκεί μάθαμε ότι υπήρχαν προβλήματα να μιλάει ως μπλοκ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταξύ βελτιώθηκε η κατάσταση και χαίρομαι που το μαθαίνω. Υπάρχει όμως μια κόποση στα Ηνωμένα Έθνη ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι τόσο δύσκολο για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαίρως να υλοποιούν. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια πάρα πολύ ατυχή στάση και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στο Συμβούλιο. Ε, στο μεταξύ έχουμε καταφέρει για κάθε θέμα χρειάζεται χωριστή απόφαση αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ή χρειάζεται άλλη ρύθμιση. Αντί δηλαδή να συντονιζόμαστε καλύτερα και να αγωνιζόμαστε για τις θέσεις μας στα Ηνωμένα Έθνη, κατάφερε το Ηνωμένο Βασίλειο να μας διχάσει. Ότι θα πρέπει πρώτα να συντονιστούμε μεταξύ μας και μετά χαιρετίσματα. Θα είναι πάρα πολύ αργά για οποιαδήποτε επιρροή. Έτσι έχει κατάσταση στα Ηνωμένα Έθνη και εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστη περίπτωση κόλληση εργίας και λυπάμαι πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλες χώρες ε, του ΟΗΕ που προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υποστήριξη και εμείς δεν μπορούμε οι ίδιοι να έχουμε θέση. Αυτό δεν ισχύει για όλα τα θέματα βεβαίως. Υπάρχουν και ζητήματα που ασκούμε επιρροή αποτελεσματικά, αλλά δεν βελτιώθηκε η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την αίτηση της Παλαιστίνης να γίνει μέλος, ε, δεν είχε προχωρήσει πολύ όταν πήγαμε η κατάσταση. Ήταν λίγο μια κατάσταση αναμονής. Οχτώ είναι τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας που θέλουν να υπερψηφίσουν την αναγνώριση της Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά χρειάζονται εννέα. Αυτό είναι το κατόφλι. Ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Προς στιγμή είναι 8 τα κράτη-μέλη και όπως γνωρίζετε τα κράτη-μέλη παραμένουν διχασμένα για το θέμα. Για την Αραβική Άνοιξη δόθηκε μεγάλη έμφαση στη ε, δημιουργία ικανοτήτων. Βεβαίως διαφορετική είναι η προσέγγιση για τη Λιβύη, δεν θα σας εκπλήξει, ή για την Τινησία, την Αλγερία ή την Αίγυπτο. Ε, σοβαρές ανησυχίες υπήρχαν ήδη από τότε για τη Συρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μάλλον η Επιτροπή Ερευνητική Συγγνώμη των Πραγμάτων ε, μιλούσε ακριβώς για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που κάνει η Συριακή κυβέρνηση. Το θέμα είναι κατά πόσο θα πρέπει η Συρία να παραπευθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αλλά δεν έχει υπογράψει το καθεστώ τη Ρώμη και αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω του Συμβουλίου Ασφαλεία και ξέρετε ότι υπάρχει ε, δυσκολία εκεί. Για τη Δυτική Σαχάρα τότε είχε θεωρηθεί ότι το κλίμα είχε χαλαρώσει μεταξύ του Μαρόκου και του μετόπου Πολυσάριο, αλλά ακόμα δεν είχε ε, οριμάσει ο χρόνος για ουσιαστική συμφωνία. Η ευθύνη για την προστασία. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη έχει γίνει πρόοδος ε, στα όργανα του ΟΗΕ, αλλά οι χώρες BRICS δυστυχώς έχουν αναπτύξει διαφορετική προσέγγιση. Ε, ευθύνη κατά τη διάρκεια της προστασίας είναι κάτι διαφορετικό. Μετά το ψήφισμα 1973 και την κρίση στη Λιβύη και την επέμβαση του ΝΑΤΟ και Αράβων και άλλων συμμάχων εκεί, η ιδέα των Βραζιλιάνων και των άλλων είναι να υπάρχει μια αυστηρή σειρά ακολουθία στην παρέμβαση ε, που αποκλείει την ταυτόχρονη χρήση διπλωματίας και βίας. Θεωρούν ότι πρέπει να ισχύει το ένα ή το άλλο. Ε, ακούστηκαν και επιφυλάξει και από εμά και από τις ΗΠΑ. Εκεί που συμφωνούμε είναι ότι η ευθύνη μας να προστατεύουμε δεν τελειώνει με το τέλος της σύραξης. Θα πρέπει να είναι και προληπτική και ανοικοδόμηση μετά το τέλος του πολέμου. Ενίσχυση κοινωνίας των πολιτών, ε, νεολαία, πολιτικά κόμματα Βέβαια για τα Ηνωμένα Έθνη αυτό είναι λίγο πιο λεπτό θέμα. Ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε πώς οι κοινοτικές προτεραιότητες εφαρμόζονται στη Νέα Υόρκη, τι δυσκολίες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, προβλέπουμε στις συστάσεις για την επόμενη Γενική Συνέλευση την 67η. Σας ευχαριστώ πολύ και αν έχετε ερωτήσεις με χαρά να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ανδρικένε μόλις κατέφτασε. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, με συγχωρείτε που καθυστέρησα, αλλά έπρεπε να λάβω το λόγο και στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Ως μέλος ε, της Επιτροπής αυτής, έλαβα μέρος στην ε, Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την 66η Γενική Συνέλευση, και μετά την ενημερώση από τον κύριο Σλαφράγκα, ήθελα να τονίσω τη σημασία την ε, συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής ΑΦΕΤ στις Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ. Θα έπρεπε να βρούμε και εναλλακτικού προορισμούς ε, στις αντιπροσωπείες μας, διότι στη Νέα Υόρκη δεν συζητήθηκαν κάποια θέματα. Θα ήταν σημαντικό να υπάρχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής ΑΦΕΤ, διότι δεν ε, συζητούνται πάντοτε μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τέτοιε συνελεύσει. Βάσει του ψηφίσματος που εγκρίναμε στι 16 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υπάρχει μια παράγραφος στην οποία προσεπρογράφω και λέει ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί απαραίτητη την αποστολή ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών μάλλον αντιπροσωπιών στις Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών. Τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, συζητήθηκαν σε όλες τις συνεδριάσεις στην Νέα Υόρκη. Οι αντιπροσωπείες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα. Νομίζω τα ανέφερε ο κ. Λάμπστορφ. Αλλά οι ειδικότερε συναντήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν με τον κύριο Σιμόνοβιτς, τον ε, Γενικό Βοηθογραμματέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του είπα προσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκείνο αντιπροσώπευε την κυρία Βιλέη, ο οποίο αναφέρθηκε σε βασικά ζητήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα από διοικητική άποψη και άποψη περιεχομένου. Μια θετική εξέλιξη που μα ανέφερε είναι ότι ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ φαίνεται να στηρίζει την θέσπιση ενό ανώτερου κλιμακίου, μια ανώτερη θέση μάλλον για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Νέα Υόρκη παρακολουθώντα ζητήματα όπω τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ακτή του Ελεφαντοστού. Βεβαίω, το Συμβούλιο και στη Γενέβη συζήτησε, συζήτησε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τον Ιούνιο του 2011 υπήρξε η δημιουργία ειδική ε, θέση για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, καθώ και ανακλήθηκε η συμμετοχή τη Λιβύη. Κάθε κράτο μέλο, λοιπόν, δέχτηκε την ε, επικριτική επικοδομητική επικριτική συζήτηση με τους ομολόγους του για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως προς την ε, Συρία υπάρχει η έκθεση της Αρμοδής Επιτροπής που μιλά για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα ήθελα να αναφέρω στους συναδέλφους, αλλά λόγω του χρονικού περιορισμού θα σταματήσω εδώ. Okay. Ευχαριστώ όλοι συνάδελφοι. Όχι, ευχαριστώ για την ενημέρωση αυτή. Και τώρα περνούμε στο τελευταίο θέμα. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Αλαφράγκα. Παρακαλώ για την αντιπροσωπεία στη Λιβύη. Πήγατε στην Τρίπολη και στη Βενγάζη, έτσι, 10 με 12 Φεβρουαρίου. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πράγματι. Πολλά μέλη της Επιτροπής μας, ο κύριος Ντανζάν, πρόεδρος της Υποεπιτροπής Άμυνας, ο κύριος Πανσέρη, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για το Μαγκρέμπ, η κυρία Γκόμες, μόνιμη συγκήτρια για τη Λιβύη, ο κύριος Κατσίν, μέλος Επιτροπής και εγώ πήγαμε στη Λιβύη 10, 11 και 12 του μηνός Φεβρουαρίου και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε αφενός τις τεράστιες προσδοκίες που δημιούργησε στον πληθυσμό η ε, εξαφάνιση του καθεστώτος του συνταγματάρχη Καντάφη και αφετέρου τις τεράστιες ανάγκες που έχει η χώρα βεβαίως. Ε, ε μπροστά λοιπόν σε αυτή την αντίφαση ε, ε, είδαμε τον πρόεδρο του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, μας είπε τι δυσκολίες έχουν και τι προβλήματα στην ασφάλεια, στην εκλογική διαδικασία που είναι καθοδόν και σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και τα μεταναστευτικά ρεύματα. Για το πρώτο θέμα συζητήσαμε και με τις μέλη της κυβέρνησης. Το βασικό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα είναι το πώς θα λύσει το θέμα της ασφάλειας και πώς οι παλιοί μαχητές θα ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις και στην αστυνομία. 150.000 είναι αυτοί η χώρα είναι ακόμα υπό τον έλεγχο των πολιτοφυλακών. Θα πρέπει να δείξει στεναρή δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει να λυθεί μια προβληματική κατάσταση. Όπως σας είπα στην αρχή, έχει να κάνει και με τα σύνορα. 4.000 χιλιόμετρα χερσαία σύνορα και 2.000 χιλιόμετρα ακτές. Λαθρεμπόριο όπλων, διακίνηση ανθρώπων. Πραγματικά είναι με μελανά χρώματα εικόνα που μπορεί κανείς να σκιαγραφή για τα προβλήματα και τη χώρα. Στείλαμε γράμμα στην κυρία Άστον και της εξηγούμε στην επιστολή αυτή λίγο τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους διάφορους μηχανισμούς και τα μέσα της για να αντιμετωπίσει αυτές ε, τις ε, ανάγκες που είναι οξύτατες. Ταυτόχρονα τα μέλη της κυβέρνησης μα διαβίβασαν και άλλες ανάγκες που έχουν ε, για από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και ανθρωπίνων πόρων και εμείς θα προτείναμε να χρησιμοποιηθούν εκείνοι οι μηχανισμοί που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το μέσο σταθερότητας, για να δώσουμε απαραίτητη και ανάλογη απάντηση. Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να αφαιρθώ λίγο και στα θέματα των εκλογών. Τον Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Η κατάσταση είναι πολύ ανισχυτική από αυτή την άποψη. Πάνω από 40 χρόνια ήταν το καθεστώς Καντάφη και ουδέποτε ε, υπήρξε προεκλογική ή εκλογική διαδικασία. Δηλαδή ο κόσμος είναι τελείως το περιθώριο της πολιτικής συνείδησης και συνειδητοποίησης για να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα ήθελα να σας πω ότι θέλουν να συνεργαστούν καταρχήν με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντίθεση με τα όσα ζήσαμε σε άλλες χώρες. Οπότε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε συνείδηση πολιτική ε, και να βοηθήσουμε τεχνικά για την εκλογική διαδικασία από τους μηχανισμούς που έχουμε θα ήταν ευπρόσδεκτη. Το νέο μέσο, η διευκόλυνση για την ε, κοινωνία των πολιτών από την πολιτική γειτονία προσφέρεται πάρα πολύ, όπως οτιδήποτε έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης. Το Euronews, για παράδειγμα, ή ε, το κανάλι του Κοινοβουλίου μας, είναι πολύ ευπρόσδεκτα γιατί πραγματικά ε, είναι στα σπάργανα όλη η προσπάθεια. ο πόλεμο γνώρισε η χώρα και έχει αφήσει πίσω του ε, σημάδια ε, και όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Θα πρέπει να καλυφθούν πάρα πολλέ ανάγκε. Είναι πάρα πολύ πενιχρά τα μέσα που έχουν στη διάθεσή του οι αρχέ του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλε αυτέ τι οξύτατε καταστάσει. Εγώ δεν θα μπω τώρα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σα είπα πώ έχει κατάσταση ασφαλεία. Οι πολιτοφυλακέ ελέγχουν ε, την κατάσταση Οι οπαδοί του Καντάφη είναι στα χέρια της, των, της ακάστοτε πολιτοφυλακής, ούτε στα δικαστήρια, ε, ούτε ε, στα χέρια του στρατού, ούτε της αστυνομίας. Ε, είναι πολύ ανισχυτική η κατάσταση και έχουμε και λαθρεμπόριο όπλων. Τέλος, Πρόεδρε, το μόνο που θα ήθελα να πω ως μήνυμα προς τα μέλη της Επιτροπής μας είναι ότι η υποδοχή που γνώρισε η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και μπορεί εδώ να συμπληρώσει κάλλιστα η κυρία Γκόμες γιατί γνωρίζει την κατάσταση της χώρας πολύ καλά. Ε, έχει πάει πανηλημένα υπό διάφορες συνθήκες και μπορεί να με συμπληρώσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπογραμμίζω ο πάρα πολύ έντονα τη θαυμάσια υποδοχή που μας επιφύλαξαν, ε, την προθυμία τους να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας είναι θαυμάσια και σπουδαία ευκαιρία και δεν θα πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη για λόγους γραφειοκρατικούς. Δεν ε, έχουν την ίδια στάση άλλοι διεθνείς ε, φορείς. Η Λιβύη για μας θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και υπό την έννοια αυτή θα ήθελα να σας πω ότι Διαβιβάσαμε τις εντυπώσεις μας στην ύπατη εκπρόσωπη για να μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Ε, είναι τεράστιες οι ανάγκες. Ήταν επιτυχής η ε, έκβαση, ε, έπεσε το καθεστώς κατάφυγα, αλλά τώρα αυτό που χρειάζεται είναι να οικοδομηθεί η χώρα να λυθούν τα υλικά προβλήματα που έχουν και να μπουν οι βάσεις για μια στοιχειώδη δημοκρατική μετάβαση που και αυτή διαφαίνεται πάρα πολύ περίπλοκη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάπως παράδοξο. Όσοι έχουν την εξουσία και τη δύναμη των όπλων πρέπει να τα παραδώσουν σε κάποιον που δεν έχει υπόσταση. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί κάποια αρχή που μπορεί να συλλέξει τα όπλα αυτά και Βεβαίω, είναι τεράστιο το καθήκον και τεράστια η αρμοδιότητα. κυρία Γκόμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πόσο εκτιμώ ότι είμαι μέλος αυτής της ομάδος και ε, ε, αναφερθώ και εις ε, τους διάφορους άλλους συναδέλφους σαν εισηγήτρια του Κοινοβουλίου που έχει πάει το Μάιο στη Βενγάζη και το Σεπτέμβριο στην Τρίπολη χαίρομαι διότι η ερμηνεία των συναδέλφων είναι η ίδια με τις δικές μου εντυπώσεις δηλαδή ότι έχουν καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα ότι θα έπρεπε η Λιβύη να αποτελέσει την πρώτη μας προτεραιότητα και αυτό όχι μόνο σαν αποτέλεσμα της επενδύσεως την οποία κάναμε τον τελευταίο χρόνο μετά από τις εξελίξεις αλλά ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα λαμβάνοντας υπόψη και τα δικά μας συμφέροντα δηλαδή ε, πρέπει να επιτύχει η κατάσταση στη Λιβύη ε, μπορεί να υπάρξει μεγάλη διαφορά και αυτό το οποίο θα επιτύχουμε εκεί αναφέρεται στα δικά μας συμφέροντα ε, σε όλους τους τομείς από πλευράς ασφαλείας η ασφάλεια της Λιβύης είναι και δικιά μας και στον οικονομικό τομέα διότι η Λιβύη είναι μια πλούσια χώρα και από πολλούς και είδαμε ότι από τις ε, χώρες της περιοχής ήταν η πιο επιδεκτική ε, να ακολουθήσει τις απόψεις μας δηλαδή με, πολλά, με πολλούς τρόπους οι Λίβοι μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι επιθυμούσαν την βοήθεια της Ευρώπης. Δεν χρειάζονται χρήματα, έχουν χρήματα. Η παραγωγή πετρελαίου επανήλθε στο επίπεδο πρώτης επανάστασης αλλά θέλουν να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους. Δεν υπήρχαν πολιτικά κόμματα, δεν υπήρχε μία ομαλή κατάσταση. Η ε, προτεραιότητα αυτής της ε, πολιτοφυλακής ε, αντιπροσωπεύει το μόνο μηχανισμό ασφαλείας στη Λιβύη διότι δεν υπάρχει πραγματικό στρατός και δεν υπάρχει πραγματική αστυνομία. Μας ζήτησαν λοιπόν ε, να βοηθήσουμε ε, και μας ζητούσαν βασικά πράγματα, ουσιώδη πράγματα, διότι πριν από μία εβδομάδα ε, ήταν 17 Φεβρουαρίου η επέτειος της Επανάστασης και ήταν πάρα πολύ αναστατωμένοι οι Λίβοι λόγω των ανακοινώσεων του ιού Καντάφη από τον ήγυρα και διότι πιστεύω ότι τώρα που ε, κατεργήθη το παλιό καθεστώς πρέπει να αποφασίζει το νέο καθεστώς ε, το οποίο είναι μεταβατικό. Ε, δεν είναι μία κυβέρνηση η οποία μπορεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις όπως παραδείγματος χάρη στο θέμα της ασφαλείας. Δηλαδή βλέπουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν αυτήν την πολιτοφυλακή και Νομίζω ότι γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαλαφράνκα. Δηλαδή με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών μπόρεσαν να εγκρίνουν τον εκλογικό νόμο που είναι πολύ σημαντικός γιατί προβλέπονται εκλογές τον Ιούνιο που δεν θα είναι τέλειες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα υπό αυτές τις συνθήκες αλλά μόνο έτσι μία κυβέρνηση θα θεωρηθεί σαν νομιμοποιημένη. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ε, παρόλο που δεν πρόκειται να υπάρχει μία τέλεια διαδικασία ε, όπως και οι διαδικασίες στην ε, Αίγυπτο δεν είναι τέλειες δεν πρέπει να τους πιέζουμε διότι γνωρίζουμε εκ προημίου ότι δεν θα είναι τέλεια η κατάσταση αλλά έτσι θα υπάρχει μια νόμιμη κυβέρνηση

και αυτές οι εκλογές εφόσον δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα ε, είναι και αυτό μία από τις δυσκολίες και είδαμε ότι 120 βουλευτές της ε, ε, συντακτικής συνέλευσης θα συνέλθουν εκ των οποίων ένα ποσοστό θα είναι από τα νέα πολιτικά κόμματα και θα πρέπει να είναι σε πλήρη ε, πλήρως ισοσκελισμένα μία γυναίκα για κάθε άντρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μία Ισλαμική χώρα όπως είναι η Λιβύη και ε, μας δείχνει ότι παρόλα αυτά υπάρχει δυνατότητα της κοινωνίας της Λιβύης να οργανωθεί παρόλες τις ατέλειές της. Οι γυναίκες ε, διαδήλωσαν ε, όταν υπήρχε στην αρχή μία ποσόστοση 10% και ε, βλέπετε ότι επέτυχαν αυτό το οποίο ήθελαν και όπως είπε και ο κύριος Αλαφράγκα αυτό είναι λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κοιτάξει να φροντίσει να έχει έναν μόνομο εκπρόσωπο να δούμε ποιες είναι οι βασικές ανάγκες τι γίνεται με την κοινωνία των πολιτών με τα μέσα εγώ βέβαια θα μπορούσα να σας μιλήσω αν είχαμε χρόνο για πολλά προβλήματα για τους φυλακισμένους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής ο κύριος Κατέιν και μετά ο κύριος Φον Λάμστορ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να παρουσιάσω έξι σημεία των παρατηρήσεών μου ο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο αντιπρόεδρος της Προεδρίας είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ρευστότητα διότι η προηγούμενη κυβέρνηση, το προηγούμενο καθεστώς αφαίρεσε ε, όλα τα έγγραφα φεύγοντας και δεν ε, έχουν ε, χρήματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν ε, προτεραιότητες που θα πρέπει να ρυθμιστούν για να ελέγχουν την κατάσταση. Και αυτό ήταν και το νόημα της ερώτησής μου σήμερα εις τον Υπουργό της Ιορδανίας. Δηλαδή, εάν η Ιορδανία θα συμβάλλει, εάν σκεφτεί κανείς ότι στην Λιβύη ε, το πρόβλημα ε, της ε, ε, της διοίκησης απλώς ε, θα βελτιωνόταν. Δεν μπορεί κανείς να βελτιώσει κάτι ανύπαρκτο, πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ο Καντάφη δεν δημιούργησε τις αναγκαίες δομές, ε, Υπήρχε μόνο, υπάρχουν μόνο οι τοπικές αρχές, οι τοπικοί φύλαρχοι και είναι μακρύς ο κατάλογος των ελλείψεων. Το τρίτο, η τρίτη μου όμως παρατήρηση είναι ότι αυτή τη στιγμή οι, οι Ορδανοί προσπαθούν να προσλάβουν και να ενσωματίσουν εις την Λιβύη πρώην στρατιωτικούς και να τους κάνουν αστυνομικούς αλλά δεν έχουν καν αστυνομικά τμήματα κτίρια δηλαδή και χρειάζεται να υπάρξει μία βασική βασική δομή της οργανώσεως κατά τρόπον ώστε η πολιτοφυλακή αυτή να μπορέσει να ενστοματωθεί στην νομική δομή διότι υπάρχει γενικό επιτελείο όχι όμως στρατός. Ε, εγώ είχα ε, διαπιστώσει αυτή την έλλειψη και εσείς κύριε Πάσκα μόνο στην ε, αεροπορία υπάρχουν επαγγελματίε στρατιωτικοί. Όχι στο στρατό ξηράς και αυτό πρέπει να αναπτυχθεί. Ε, έχουν πρόβλημα και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις διότι οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων αναρωτήθηκαν ε, η δημοκρατία είναι αυτή, υπάρχει καταπίεση ε, φοβούνται πρώτων εκλογών διότι οι, αυτοί που θα εκλεγούν θα υποστηρίξουν τις δικές τους φυλές. Δεν έχουν τις βασικές αρχές τις οποίες εμείς έχουμε στερνιστεί για να λειτουργήσουμε σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Και γι' αυτό έκανα και τις ερωτήσεις μου στον εκπρόσωπο της Ιορδανίας. Ο νεότερος, ο, νεότερος ο οποίος έχει ζήσει εκλογές είναι 70 χρονών τώρα διότι ε, έχουν περάσει 40 χρόνια δικτατορίας. Ως εκ τούτου είναι πολύ ε, ηλικιωμένοι αυτοί που έχουν ξαναζήσει εκλογές. Υπάρχουν ε, διάφοροι πολιτισμοί, διάφορες θρησκείες στη Λιβύη. Πολλοί δεν μιλούν την αραβική γλώσσα και είναι αποκομμένοι τελείως από τα τεκτενότητα φαινόμενα στην ε, Λιβύη και είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Ξέχασα και δύο άλλα σημεία. Καταρχήν τον ρόλο που ανέφερε ο συνάδελφος Φράνκα, δηλαδή τι μπορούμε εμείς να κάνουμε. Η κοινοβουλευτική μας τηλεόραση μπορεί να ετοιμάσει διάφορα σποτ τα οποία θα μπορέσουν να διευκρινίσουν και να προβληθούν οι ε, εξηγώντα την ε, κοινοβουλευτική δημοκρατία ε, ότι ήταν θετική στις προτάσεις της ε, κάθε και η σημερινή συζήτηση σε αυτό αποβλέπει να μπορέσει να κινητοποιηθεί και το Προεδρείο του Κοινοβουλίου άπαξ και θα γνωρίζουμε πόσες μεγάλες είναι, πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες δηλαδή η, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρει εκτιμήσεως και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε ε, ε, θετικά. Και ε, η Λιβύη έχει ε, μεγάλες δυνατότητες οι οποίες έχουν παραγνωριστεί. Η Λιβύη επιπλέον δεν είναι μόνο η Τρίπολη, η οικονομία της Λιβύης είναι στη Βενγάζη και η πνευματική άρχουσα τάξη είναι στην Βενγάζη και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανωθεί καλύτερα, να ανοίξει ένα γραφείο και στη Βενγάζη. Το σκεφτήκαμε γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο της Λιβύης Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό ενιαίο προξενείο κατά τρόπον ώστε όλες οι χώρες να μπορούν να εκδίδουν θεωρήσεις και να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να ταξιδεύσουν 350 χιλιόμετρα μέχρι την Τρίφολη εφόσον πρόκειται για βιομετρικά έγγραφα και ολόκληρη η οικογένεια θα πρέπει διαφορετικά να ταξιδεύει μέχρι την Τρίπολη και πίσω. Δύο φορές μάλιστα, όχι μία. Λοιπόν, ένα τέτοιο προξενείο θα μπορούσε να είναι κάτι νέο, κάτι πολύ θετικό, κάτι πολύ ορθολογιστικό και θα μπορούσε να έχει και μεγάλη απήχηση. εγώ δεν, το, δεν σκόπευα να, να πω κάτι τέτοιο, αλλά τώρα μου ήρθε η ιδέα και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό, αλλά ε, για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο, στο Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχω να κάνω μία σύντομη ερώτηση στον Ιγνάσιο. Πήγε στη Τρίπολη, μπορεί κανείς να ταξιδεύει εκτός της Τρίπολης ε, με την ε, αποστολή. Υπάρχουν α, α, οι είναι δυνάμεις ασφαλείας ή απλώς ο, λαιλατούν. Πάρα πολύ γρήγορα, κύριο Σαλαφράγκα η Υπηρεσία εξωτερική Δράσης μα είπε ότι έπρεπε να έχουμε ένα κήτα ασφαλεία ε, που ήταν ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο και ε, ένα κράνος. Ευτυχώς δεν τους δώσαμε σημασία και ε, κυκλοφορήσαμε ελεύθερα με καλή ασφάλεια. Αλλά όπως είπε πολύ ωραία ο κύριος Κατσίν δεν υπάρχει στρατός ούτε αστυνομία ε, είχαμε δείπνο με την Υπουργό Υγείας ε, μόλις καταφέραμε να φύγουμε από το μπούνκερ του ξενοδοχείου και επιστρέφοντας στο αυτοκίνητό της, τις επιτέθηκαν. Ε, κάποιοι από πολιτοφυλακή είναι στο έλεος των πολιτοφυλακών. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει ε, αστυνομία που να συλλαμβάνει κάποιους και να τους προσάγει στη δικαιοσύνη. Εγώ πήγα μόνο στην Τρίπολη, δεν είχα χρόνο να πάω αλλού. Είχα ένα ε, αστυνομικό που με συνόδευε ένα μικρό κύριο που ήλεγχε όλο το αεροδρόμιο, αλλά ήταν και αυτό στα χέρια των πολιτοφυλακών. Τι να κάνουμε, έτσι έχει κατάσταση σήμερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος. Ελπίζω αν είναι κοντή και μικρό να έχουν μεγάλα όπλα τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ όλους σας ε, για τη συνεργασία. Πριν φύγουμε όμως θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 20 Δεκεμβρίου του 2011. Διαφωνεί κανείς? Ωραία, εγκρίνουν τα πρακτικά. Ε, λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 9 ακριβώς έχουμε ψηφοφορίες. Ακριβώς όμως και να φέρετε και τις κάρτες σας γιατί ψηφίζουμε στις 9.